Liebe Kolleginnen, liebe Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρω ότι έχετε και εσείς όρεξη να μην μείνετε εδώ μέχρι αργά το βράδυ και γυρίσετε στα δωμάτια σας. Ξεκινάμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής του Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Την ημερήσια διάταξη την έχετε λάβει. Ε, δεν έχω λάβει εγώ από πλευράς μου. Εγκρίνεται λοιπόν η μερίσια διάταξη έχετε, θε, ε, γλώσσες επίσης έχετε ενημερωθεί ποιες είναι. Έχουμε και web streaming και ξεκινώ με την ημερήσια διάταξη στο σημείο 3. Διαπραγματεύσεις τριμερούς διαλόγου. Ο Ρίτσαρτ Ashworth, ο εισηγητής, καλό θα ήταν να ήταν εδώ βέβαια σε αυτό το σημείο. Αλλά πού είναι. Έτσι λοιπόν, μήπως να δούμε πρώτα το σημείο 4 γιατί ο κύριος Βον είναι εδώ. Καλή ιδέα, καλή ιδέα πρόεδρε. Καλώς. Επομένως πάμε στο σημείο 4 Τι δίνω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαρίστω ε, να συζητήσουμε πρώτα το δικό μου θέμα. Βέβαια δεν είναι ε, η πρώτη συζήτηση που έχουμε για την ε, το πρόγραμμα εγγύησης για τους νέους. Είμαι ευτυχής που σήμερα έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για αυτό το σημαντικό θέμα. Από την τελευταία μας συζήτηση έχω συντάξει την έκθεση και στη συνέχεια έλαβα 79 τροπολογίες που κατέθεσαν οι διάφοροι συνάδελφοι και για την ώρα προσπαθώ να δω κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να συντάξουμε κάποιες συμβιβαστικέ τροπολογίες ώστε να καλύψουμε κάποιες από αυτές τις 79 που υπέβαλαν οι συνάδελφοι. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από τους συναδέλφους. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους και ιδιαίτερα τον ε, Λαφράγκα Σάντσες Νιέρα που δεν νομίζω ότι είναι εδώ αλλά εντυπωσιάστηκα από την ε, τροπολογία του 17. Συνάδελφοι δείτε τι είναι που ενημερώνει κάποια από τα νούμερα που αφορούν την, ε, τα ποσοστά ανεργίας νέων σε ολόκληρη την Ένωση, αλλά και κάποια στοιχεία που σχετίζονται με τον αριθμό των νέων που έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα εγγύησης για τους νέους. Κάθε τροπολογία είναι φυσικά ευπρόσδεκτη, αλλά αυτή όλος ιδιαιτέρως ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Όταν διαβάζω ε, όλες τις ε, τροπολογίες ε, έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι θεώρησαν πως επιπλέον χρηματοδότηση θα χρειαζόταν αυτό το πρόγραμμα αλλά επίσης πολλοί εκ των συναδέλφων τόνισαν ότι οι εθνικές κυβερνήσεις Ε, χρησιμοποιούν και δικούς τους πόρους για να κατοπολεμήσουν την ανεργία των νέων. Κάτι ακόμα σημαντικό είναι ότι γνωρίζετε πως το πρόγραμμα εγγύησης για τους νέους ξεκίνησε πολύ αργά για πολλούς και διάφορους λόγους, ωστόσο έχει σημειωθεί πρόοδος τώρα, αλλά βεβαίως περισσότερα ακόμα θα πρέπει να γίνουν. Και ιδιαίτερα συνάδελφοι μέσω των τροπολογιών τους τόνισαν ότι θα πρέπει να διευρυνθεί αυτό το πρόγραμμα γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί νέοι που δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδου προγράμματα. Γι' αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί. Κάποιε τροπολογίε όσον αφορά την ποιότητα. Όταν είχαμε την προηγούμενη ανταλλαγή απόψε, εγώ και ορισμένοι άλλοι παρατηρήσαμε ότι είναι καλό να έχουμε σχέδια για την εγγύηση για του νέου, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι είναι και ποιοτικά. Στο παρελθόν, α πούμε, στο Ηνωμένο Βασίλειο συχνά είχαμε προγράμματα για τους νέους, όπου οι νέοι έπρεπε να δουλέψουν, έπρεπε να φτιάξουν ε, καφέ, να κάνουν φωτοαντίγραφα κτλ. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό για να εξασφαλίσουμε ότι όντω ε, είναι ποιοτικέ οι θέσει απασχόληση που προσφέρουμε. Στην προηγούμενη λοιπόν ανταλλαγή απόψεων ε, τονίστηκε το θέμα τη ανάγκη για ποιοτικέ θέσει απασχόληση, αλλά θα πρέπει να ορίσουμε και την ποιότητα. Τι εννοούμε όταν λέμε για ποιοτικέ θέσει απασχόληση απασχόλησης. Στο κείμενο λοιπόν Έχουμε τώρα μια πρόταση για το τι θα μπορούσε να είναι ο ορισμός αυτός και χρησιμοποιούμε ότι ε, ε, λαμβάνει υπόψη το, το ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τις μαθητείες αλλά και για τους κοινωνικούς εταίρους ε, όσον αφορά το πλαίσιο των μαθητιών και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για έναν ορισμό. Εγώ και άλλοι συνάδελφοι, όπως η Χάιντερ, Έχουμε καταθέσει τροπολογίες ε, για να πούμε τι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον ορισμό των ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Πρέπει να το συζητήσουμε νομίζω γιατί έχουν κατατεθεί διάφορες τροπολογίες που προσπαθούν να ορίσουν ε, τι σημαίνει ε, ποιοτική προσφορά. Κάποιοι συνάδελφοι επίσης έχουν ε, ονοματίσει ε, κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν ε, όπως θα έπρεπε αρκετά γρήγορα το πρόγραμμα για την εγγύηση για τους νέους. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές όσον αφορά αυτή την τακτική του να δαχτυλοδείξουμε και να παραδειγματίσουμε τα κράτη-μέλη που δεν το εφαρμόζουν. Καλύτερα είναι να τονίσουμε συστημικά ζητήματα και να μην δαχτυλοδείξουμε κράτη-μέλη κατά τη γνώμη μας, αλλά ίσως είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε απόψε ή σε κάποια άλλη στιγμή. Τέλος, Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι την εβδομάδα 18 ε, Σεπτεμβρίου θα γίνει μια συνάντηση των συντονιστών για να συζητήσουμε τις τροπολογίες και φυσικά και οι σκιώδεις θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουμε τις τροπολογίες και ε, τις συμβιβαστικές. Ο κύριος Αλαφράγκα μόλις ήρθε, ανέφερα προηγουμένως, ε, Νάσια πολύ εκτιμώ την ε, τροπολογία σου υπαριθμών 17 που ενημερώνει τα στοιχεία για τους νέους άνεργους. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Δεν στήκανε το λόγο από ό,τι βλέπω. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το θέμα της μερικής διάταξης. Πάμε στις ψηφοφορίες. για τις 25 Σεπτεμβρίου, στις Βρυξέλλες δηλαδή. Επανέρχομαι στο σημείο 3, καλώς ορίζοντας και τα μέλη της Επιτροπής των Προϋπολογισμών. Έκθεση για τις συνεδριάσεις του τριμερούς διαλόγου για το δημοσιονομικό κανονισμό. Τρίτη συνεδρίαση σήμερα. Καλώς ορίζω τους συναδέλφους λοιπόν της Επιτροπής των Προπολογισμών. Είμαι και εκ μέρους της Επιτροπής των Προπολογισμών εισηγήτρια. Έχουμε συνεισηγητή τώρα από πλευρά της Επιτροπής Ελέγχου των Προπολογισμών, τον Ρίτσαρντ Άσχουρθ και του δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε μπορώ να πω. Στην ε, μεικτή επιτροπή που έχουμε είχαμε δύο συνεδριάσεις τριμερούς ε, διαλόγους αρχίζοντας 29 Αυγούστου και στις 30 που συζητήσαμε τους κανονισμούς τους ε, δημοσιονομικούς και προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερη πρόεδρο, να δούμε ποια ήταν τα θέματα τα οποία ήταν επίμαχα. Θα έπρεπε να πω ευθύ εξ αρχής ότι έπρεπε να συμπληρώσουμε αυτή την εργασία, να την ολοκληρώσουμε το φθινόπωρο, κατά προτίμηση το τέλος Οκτωβρίου. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ε, μετά από 10 ε, συνεδριάσεις είχαμε, ε, ασχοληθήκαμε με 60 άρθρα, εδώ έχουμε 280 άρθρα και ελπίζω ότι μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε καλύψει ακόμα 40. Είναι βεβαίως πάρα πολύ μεγάλη μακρόπνοη εργασία και θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην την, ΑΣΜΑ που έκανε πάρα πολύ καλή εργασία και σε όλους τους συνεργάτες μου. Υπάρχουν μερικά θέματα τα οποία συμφωνήσαμε με τους θεσμούς. Υπάρχουν θέματα όπου είχαμε ε, συμφωνία ως προς την διατύπωση, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν ε, μερικές, μερικά βασικά θέματα, ουσιαστικά θέματα, όπου δεν έχουμε καμία συμφωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν, κυρίως με το Συμβούλιο. Γι' αυτό τα αναβάλαμε για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στα θέματα αυτά, τα ουσιαστικά να επανέλθουμε και να τα συζητήσουμε αργότερα. Νομίζω ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχουν δύο σημεία που θα ήθελα να θέσω ε, ε, σχετικά με τον χρονοδιάγραμμα Νομίζω ότι πάντοτε διευκρινίσαμε από την αρχή ότι ήταν φιλόδοξο ε, να τελειώσουμε την εργασία αυτή τόσο σύντομα και αυτό αποδεικνύεται ότι είναι δύσκολο. Και βεβαίως δεν είμαι ικανοποιημένο από την αντίδραση, από την δράση, από την Επιτροπή ε, στις αναφορές που μας κάνει ε, δίνοντάς μας ένα σχόλιο, μια συμφωνία, μια αντίδραση τα τρία μέρη βεβαίως θα βρεθούμε στο ίδιο σημείο όταν επανέλθουμε. Πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση για να προδέψουμε καλύτερα στο μέλλον. Εν τω μεταξύ, έχουμε θέματα τα οποία αναφέρουμε στους σκιώδεις ε, και έχουμε μερικά θέματα τα οποία παραπέμφθηκαν έτσι και Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ακόμα πάρα πολλή εργασία να κάνουμε και θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την εργασία αυτή μέχρι το τέλος του έτους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να συμπληρώσω εδώ ότι έχουμε περισσότερα εκκρεμή ζητήματα από ζητήματα στα οποία έχουμε συμφωνήσει. για τους εκπροσώπους της Επιτροπής αλλά και των κρατών μελών θα ήταν καλό να συμπληρωθεί με την περαιτέρω εργασία όπως αναφέρεται άλλωστε το σύνολο των ε, εκκρεμών σημείων για τα οποία έχουμε πει ότι πρέπει να γίνει περαιτέρω δουλειά. Έχουμε ένα περιθώριο μέχρι τον Οκτώβριο, αλλά το αποθυματικό κρίσος, ε, τα εμβάσματα, το carryover, προθεσμίες, όλα είναι κρεμή. Και αρκετά δύσκολα ζητήματα. Εμείς πάντως θα αγωνιστούμε για να διαφυλάξουμε και τις προνομίες του Κοινοβουλίου. Άρθρα 2, 12, 13, 14, 15, 17, 24, 27 έως 30, 31 έως 34, 35, 36, 39, 42, 43, 51, 60, 61, 59. Όλα αυτά για να σας δώσω μια εικόνα της δουλειάς που μένει ακόμα να γίνει. Αυτά έχουμε να πούμε εμείς. Έχετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια για τον τριμερή διάλογο. Όχι. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Είχαμε προβλέψει όμως ε, ψηφοφορίες για τις 8 και 4. Θα μπορούσαμε και τώρα να ψηφίσουμε βέβαια, αν θεωρείτε ότι είναι μου. Κανονισμός Eurojust. αν θεωρείτε ότι οι ομάδες είναι σε θέση να προχωρήσουν την ψηφοφορία. Κανονισμός Eurojust. Σημείο 5 στην ημερήσια διάταξη. Γιατί το 4 το συζητήσαμε νωρίτερα. Παρακαλώ να βγάλετε τις κάρτες σας για την ψηφοφορία. Γνωμοδότηση. Για την Επιτροπή των Εσωτερικών Υποθέσεων. 130 και είναι οι τροπολογίες μας. Ξεκινώ. 42. Υπέρ κατά. Αποχές απερίφθη, 43 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 44 είχε καλυφθεί, 45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 46 υπέρ, κατά αποχές, να απολυθεύσουμε, 46. 46. Πέρας. Εγκρίνεται. Α, όχι, με συγχωρείτε, δεν το βλέπω καλά από εδώ που είμαι. Απερίφθη. Με συγχωρείτε. Δεν είχα καλή οπτική γωνία. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 49 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 50 σε τμήματα με προφορική τροπολογία, δεν βλέπω αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, καλύπτονται και 51-52, 53 τώρα υπέρ, κατά αποχές απερίφθη, 54 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 55 υπέρ, κατά περίφθη, 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε παρακαλώ το 3 πέρας εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 58 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 59 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 60 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 61 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 62 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 63 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 64 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 65 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 η 66 πρέπει να ψηφιστεί τώρα γιατί έχει καλυφθεί τμήματα το πρώτο τμήμα της 66 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απερίφθη δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 σε δύο τμήματα το πρώτο παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απερίφθη 60 η 68 έχει καταπέσει 69 δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές απερίφθη δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 Ωραία, υπέρ, κατά αποχές απερίφθησαν. 11 υπέρ, κατά αποχές ε, εγκρίνεται, καταπίπτει 87, στην 88 τώρα υπέρ, κατά αποχές απερίφθη και πάμε στην 89 έως 96 με μια ψηφοφορία ομού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται η 12 κατά πίπτη όχι δεν καταπίπτει 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, πρέπει να έχει καταπέσει. Α, ναι, με συγχωρείτε, λέει η Πρόεδρος. Και πάμε στην 97 που επίσης έχει καλυφθεί. 98 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 99 δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102-103 έχουν γλωσσικό χαρακτήρα μόνο 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 106 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 110, 111, 112 με, σε μια ψηφοφορία παρακαλώ υπέρ κατά αποχές ε, απερίφθησαν, 113 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 115 υπέρ κατά αποχές 115 παρακαλώ να επελθέψουμε. 115 ολοκληρώνεται η ψηφοφορία και απερίφθη. 116 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 117 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 118 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 122 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 123 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 ε, υπέρ κατά αποχές απερίφθη 21 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 22 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές ε, απερίφθη 26 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 29 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 32 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 33 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 34 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 35 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε την 35. Πέρας. Απεριφθεί 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 37 υπέρ κατά αποχές Απεριφθεί 38 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 39 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 40 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 41 υπέρ κατά αποχές και απερίφθη και έτσι έχουμε φτάσει στο σύνολο της ψηφοφορίας για τη γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε αρχής ψηφοφορία. Όχι, μυστική ψηφοφορία δεν πρέπει να είναι. Εντάξει, το μαθαίνουμε σιγά σιγά. Παρακαλώ λοιπόν για άλλη μια φορά να επαναληφθεί η τελική ψηφοφορία. Κάποια κάρτα μένει ακόμα μυστική, δεν φαίνεται. Όχι, εντάξει, 15 υπέρ, μία ψήφος κατά. Σα ευχαριστώ πολύ. Για να καταλάβουν οι πάντες τι κάναμε τώρα. Είναι πολύ σημαντικό το, το τι έγινε έτσι η ψηφοφορία τώρα για να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του νέου ευρωπαϊκού τοπίου στον τομέα της εφαρμογής του δικαίου. Γιατί είχαμε δύο δυνατότητες, είτε ζητούμε από τα κράτη-μέλη να το αναλάβουν, όπως το μέχρι τώρα που δεν συνέβαινε τίποτα, είτε αναθέτουμε στην ευρωπαϊκή, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Νομική Επιτροπή με την έγκριση μια σειρά τροπολογιών De Jong έχει επιλέξει τη διακυβερνητική οδό που δεν ήταν καθόλου σωστή. Εγώ χαίρομαι που στη δική μας ε, ε, γνωμοδότηση κάναμε τις επιλογές που κάναμε. Έχω μιλήσει και με τον συνομιλητή. Είμαι πολύ περήφανη για αυτό που κάναμε. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να έχει ένα ρόλο ισχυρό, σοβαρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις ε, εκθέσεις της Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών όπως έχει συμβεί μέχρι τώρα και καλό θα ήταν να μην αποκλειστεί στο επόμενο αυτό βήμα. Αυτό για τις μεγάλες γραμμές. Όταν ξέρετε ότι στις, οι συνεδριάσεις της Eurojust ούτε καν κοινοποιούν τις ε, συνεδριάσεις, τις ημερήσεις διατάξεις. Ε, στην Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών όταν γίνονται αυτές οι συναντήσεις ε, με την ηγεσία του Eurojust. Ε, ούτε καν με διάταξη δεν μπορούμε να δούμε. Γι' αυτό λοιπόν το έχουμε συμπεριλάβει και ελπίζουμε ότι η Επιτροπή εσωτερική Πολιτικής Ιστορικών θα αλλάξει γνώμη στην υπόθεση αυτή. Έχω συνομιλήσει και με τον εισηγητή όπως είπα γιατί δεν μπορούμε να έχουμε εδώ ουσιαστική ευρωπαϊκή συνεργασία στην οποία η δική μας Επιτροπή πάντοτε επιμένει. Αυτά. Μας έχουν μείνει περίπου 30 λεπτά μέχρι να έρθει ο Επίτροπος Χάν. Μπαρτ. Να δούμε την απαλλαγή. Το δικό σου κομμάτι, Συμβούλιο Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω όντως ότι ότι θα έχουμε μια άσκηση πολύ εύκολη για αυτήν την απαλλαγή. Ξέρετε όλοι το πλαίσιο ε, σχετικά με το σημείο αυτό. Αναβάλαμε για τον Αυρίλιο την απαλλαγή μετά από τόσες φορές και τόσες επαναλήψεις, αλλά με ένα πλαίσιο κάπως διαφορετικό. Ε, πρόεδρος της Επιτροπής και εγώ είχαμε επαφές με το Συμβούλιο και το Συμβούλιο μας κάλεσε να κάνουμε μια πρόταση non-paper. Δηλαδή να συντάξουμε ένα έγγραφο, ένα non-paper το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο ε, για την απαλλαγή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν. Είναι σαφές ότι το Κοινοβούλιο χορηγεί την απαλλαγή, το Συμβούλιο γνωμοδοτεί σχετικά με τη χορήγηση αυτής της απαλλαγής. Εκεί όπου τα πράγματα δυσκολεύουν είναι ότι δεν υπάρχει καμία ανταλλαγή πληροφοριών. Εφόσον δεν απαντούν στις ερωτήσεις μας, ενώ τα άλλα θεσμικά όργανα απαντούν στις ερωτήσεις μας. Εργάστηκα λοιπόν μετά την συζήτηση για την απαλλαγή τον μήνα Απρίλιο και μετά την ψηφοφορία τον μήνα Απρίλιο στην Ολομέλεια, εργάστηκα με τον Σκιώδη εισηγητή και είχα ε, μια πολύ καλή υποστήριξη από την γραμματεία και θέλω αυτό να το τονίσω. Εργαστήκαμε για μια πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα non-paper όπου κάνουμε προτάσεις στο Συμβούλιο για να ρυθμίσουμε ορισμένα προβλήματα. Η άσκηση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είχαμε τρεις συνεδριάσεις, είχαμε μια διαβούλευση η οποία ήταν πολύ επικοδομητική και με όλες τις ομάδες τελικά καταλήξαμε σε ένα κείμενο ε, το οποίο συμφωνήθηκε. Το κείμενο αυτό υποβλήθηκε και στους συντονιστές της Επιτροπής μας. Και τώρα υπάρχουμε λοιπόν μια πρόταση κειμένου. Τι να κάνουμε τώρα, τι κάνουμε και αυτό είναι ένα ερώτημα που απευθύνω στους συντονιστές όλων των πολιτικών ομάδων. Θα έπρεπε το κείμενο αυτό που θα προτείνει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου ε, και που εγκρίθηκε από τους συντονιστές θα πρέπει το κείμενο αυτό να υποβληθεί στην διάσκεψη των Προέδρων και στους επικεφαλείς όλων των πολιτικών ομάδων. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από όλους τους συντονιστές να ασκήσουν ε, πίεση πάνω ε, στους Προέδρους των πολιτικών ομάδων για να επικυροποιήσουμε το θέμα αυτό και να το ρυθμίσουμε τον, αυτό το μήνα, διότι μόνο από τότε το κείμενο θα μπορέσει να αποσταλεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συμφωνία της διάσκεψης των Προέδρων για να σταλεί επίσημα στο Συμβούλιο. Εν τω μεταξύ, και εγώ, η Πρόεδρος και εγώ, η Συγητής, θα μπορούσαμε να έχουμε μια πρώτη άτυπη επαφή με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου για να δούμε ε, ποια είναι η κατάσταση για ε, να δούμε αν το Συμβούλιο θα υποβάλει το κείμενο αυτό ε, στο Κοροπέρ για να δούμε μετά από χρόνια σύγκρουσης θα μπορέσουμε να, να διευκρινίσουμε τα θέματα και να έχουμε ομελές σχέσεις ανάμεσα σε δύο θεσμικά όργανα που σέβονται τις συνθήκες όπου είμαστε όλοι όριμοι και ενήλικες και όπου πρέπει να γίνει σεβαστό το δικαίωμα στην πληροφόρηση. Αυτό είναι το ιστορικό, το πλαίσιο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα υποβάλλω την έκθεσή μου. Όλα αυτά δεν έχουν ακόμα επικυρωθεί. Δεν μπορώ λοιπόν να σας ε, συστήσω να δώσετε απαλλαγή στο Συμβούλιο και το σχέδιο εκθεσής μου αφήνει ακόμα πολλά εκκρεμή θέματα. Το θέμα της χορήγησης της απαλλαγής εκκρεμή. Η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι εάν το non-paper γίνει δεκτό από το Συμβούλιο, θα είναι η απαλλαγή ε, για του χρόνου που θα είναι καθοριστική. Θα δούμε αν θα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αυτό λοιπόν που έκανα για την έκθεση, έγραψα ορισμένες διατάξεις για να πω στο, στο Συμβούλιο ότι εκτιμούμε ορισμένα πράγματα το Συμβούλιο είναι λίγο πιο διαθέσιμο και διατεθειμένο να ανταλλάξει ορισμένες πληροφορίες. Αλλά παρόλα αυτά λέω ότι για την απαλλαγή 2015 υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Δεν το αναπτύσσω αυτό ενδελεχώς σήμερα το βράδυ. Όλοι μπορείτε να διαβάσετε το κείμενό μου, την έκθεσή μου, αλλά θα σας παρουσιάσω μερικά σημεία. Η παράγραφος 6 της δεύτερης έκθεσής μου επισύρει την προσοχή πάνω σε μια πραγματική βελτίωση στις σχέσεις με το Συμβούλιο, διότι για πρώτη φορά το Συμβούλιο έστειλε στο Κοινοβούλιο τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, τις Annual Activity Reports. Αναφέρω επίσης αυτό το non-paper το οποίο σας παρουσίασα στη δεύτερη εκθεσή μου. Λέω ότι κάνουμε αυτήν την άσκηση και θα στείλουμε το κείμενο αυτό, το λέω στην παράγραφο 7, στην διάσκεψη των Προέδρων. Επίσης επισύρω την προσοχή σας στην παράγραφο 11, όπου από τη μια αφενός λέμε κάτι το θετικό στην πρώτο μέρος της παραγράφου ότι το 2015 δημοσιεύτηκαν νέες κατευθυντήριες γραμμές διοντολογίας για το Συμβούλιο και μετά κάποια επιφύλαξη, κάτι το αρνητικό. Εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι οι κανόνες του Συμβουλίου σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών εξακολουθούν να μην είναι ε, δημόσιοι κανόνες διαθέσιμοι στο, στο κοινό, κυρίως σχετικά ε, με τους καταγγέλτες. Επίσης δεν υπάρχει μητρό διαφάνειας και στην παράγραφο 12 και στην παράγραφο 13 ζητώ από το Συμβούλιο να εκπονήσει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές κατά της διαφθοράς και επίσης περισσότερη ανεξαρτησία στις ίδιες τις δομές του Συμβουλίου. Μετά υπάρχει και η παραγραφός 18, όπου και πάλι κατακρίνω το Συμβούλιο εφόσον ε, λυπούμε επειδή το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην απαντά στις ερωτήσεις, στις γραπτές του Κοινοβουλίου. Αλλά, το επαναλαμβάνω, εάν το, κοινοβούλιο, το Συμβούλιο με συγχωρείτε, μπορεί να δεχθεί το non-paper και να το υποβάλει στο Κορεπέρ, θα έχουμε κάνει ένα βήμα προόδου και θα μπορούμε να έχουμε ομαλές σχέσεις με το Συμβούλιο για την απαλλαγή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ελπίζω η άσκηση αυτή να είναι θετική και να στεφτεί με επιτυχία. Ξέρω πολύ καλά ότι το να είναι κανείς εισηγητής για την απαλλαγή του Συμβουλίου δεν είναι κάτι το εύκολο, διότι οι σχέσεις είναι κακές και αν κατορθώσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα, να ε, υπερνικήσουμε το εμπόδιο, θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειες, για τη στράτευση. Θα προσπαθήσουμε βεβαίως να τηρήσουμε και τα χρονοδιαγράμματα. Πάει στη διάσκεψη των Προέδρων σήμερα και θα δούμε από εκεί τι θα προκύψει. Στιχόφσκι τώρα και μετά η Αλασέντερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική παρουσίαση του θέματος. Είμαι βέβαιος ότι έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος σε αυτό το τομέα και είμαι ευτυχής που μετά ε, τρία χρόνια μπορώ να πω ότι οι σχέσεις μας με το Συμβούλιο που ήταν πολύ άσχημες έχουν σημειώσει πρόοδο. Παράγραφοι 7 και 11 πιστεύω είναι ε, μία πρόοδος, αλλά μέχρι ότου να έχουμε μια συμφωνία που να είναι συγκεκριμένη, δεν θα έχουμε λόγο για να χαρούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι διαφανής η διαδικασία. Και όσον μας αφορά χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, προβλήματα με το νέο κτίριο που κατασκευάζεται, αλλά ε, ο προϋπολογισμός αυξήθηκε πολλές φορές, ακόμα και η Ίγκη προσπάθησε να βρει το πραγματικό κόστος ε, για αυτό το κτίριο για και το επιπλέον που προσθέθηκε προσθέθηκε όλη, τη, όλη την ώρα και ακόμα δεν έχουμε πάρει ξεκάθαρη απάντηση. Ε, πιστεύω πως πρέπει το Συμβούλιο να μας ενημερώσει για αυτά τα σημαντικά θέματα γιατί οποτεδήποτε υπάρχουν ε, προβλήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε αφορούν ε, τα κτίρια, το κτίριο της, ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρέπει να είμαστε στη θέση να εξηγήσουμε στους ψηφοφόρους μας ποιο είναι το κόστος της Ένωσης. Αυτά. Κύριε Ιαρασέντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Στάες για την μεγάλη του προσπάθεια και για τα... για το περίπλοκο αυτό θέμα δεν θέλουμε να χάσουμε ε, τις δυνατότητές μας γιατί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα παρά το γεγονός ότι ε, πρόκειται για τέτοια θέματα που αφορούν περισσότερο το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο έχει πάντα από μόνο του ε, το πράσινο φως. Θα πρέπει λοιπόν η έκθεση αυτή να, ε, να αφήσει ανοιχτή, ανοιχτό το ζήτημα του κατά πόσο θα δώσουμε ή όχι την απαλλαγή για να δούμε αν κατά τη γνώμη του το Συμβούλιο έχει οριμάσει ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε την απαλλαγή αυτή την επόμενη χρονιά. Για να μπορέσουμε δηλαδή να καταφέρουμε να αλλάξουν τα πράγματα, να δούμε αν υπάρχει καλή βούληση από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να το δούμε ξεκάθαρο. Ο Γενικός Γραμματέας που ήταν ο εκπρόσωπος της Προεδρίας φάνηκε να είναι έτοιμος να απαντήσει στα διάφορα ερωτήματα στη διάρκεια του έτους, έδειξε καλή θέληση, όμως τελικά αυτό που θέλω να ζητήσουμε από τον ε, κύριο Στάση να μας πει αν τελικά πιστεύει πως ε, πραγματικά μπορούμε με βάση την ε, εργασία που κάνει να έχουμε μια σαφή ένδειξη για το αν θα πρέπει να υπερψηφίσουμε ή όχι την απαλλαγή. Εγώ αυτό ήθελα να ξέρω. Έχουμε όλοι δείξει καλή βούληση, όλοι έχουμε φέρει εδώ βελτιώσεις, αλλά που δεν γίνονταν δεχτές. Ίσως τώρα να έχει αλλάξει η κατάσταση, όχι τόσο ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αλλά σε αυτή την Επιτροπή για άλλους λόγους. Και αυτό θέλω να δω με τον κύριο Στάις, να, να καταλάβω τι θα γίνει τελικά. Γιατί διαφορετικά επικρατεί μια σύγχυση που θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα βελτιώσει. Ähm, Άρα το θέμα της αναγνώρισης καλής πίστης το βλέπουμε συχνά μαζί με την αυθαιρεσία. Κύριο Στάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι το μόνο συγκεκριμένο ερώτημα που τέθηκε είναι της Ίνες. Θα προσπαθήσω να απαντήσω, πρέπει εξάλλου να απαντήσω, διότι διάβασα σήμερα το πρωί ότι ήταν η 7η Ευρωβουλευτής, η πιο επιδραστική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το Human Watch. Συγχαρητήρια, Ίνες εβδόμη μεταξύ των βουλευτών που είναι πιο επιδραστική. Νομίζω ότι η απάντησή μου θα είναι σαφής. Η, καλή θέληση δεν αρκεί, δεν θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε. Υπάρχει καλή θέληση, την έχουμε και νομίζω ότι από την πλευρά μας κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Αυτό το non-paper συντάχθηκε και χαίρομαι που άκουσα από την Ίνες ότι η επιστολή θα πάει στην διάσκεψη των Προέδρων Ήρθε λοιπόν η στιγμή να επισπεύσουμε και να ζητήσουμε από τους Προέδρους των πολιτικών ομάδων να κάνουν τη δουλειά τους για να μπορέσουμε να πούμε αυτή είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον τρόπο εργασίας του Συμβουλίου για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο για την απαλλαγή. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε αυτή την άτυπη συνεδρίαση με την Πρόεδρό μας και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε ε, ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου, να δούμε αν είναι ε, μια λύση που θα μπορούσε να υιοθετήσει το Συμβούλιο, διότι για την ώρα δεν είμαι βέβαιος και θα πρέπει να δούμε ε, ποια είναι η κατάσταση. Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε για την ώρα, για την απαλλαγή 2015 αυτή καθεαυτή, νομίζω είναι ότι πρέπει να εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε τη θέση που έχουμε από το Σεπτέμβριο και ακόμα για περισσότερο χρόνο. Δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες, θα τους πούμε, για να σας χορηγήσουμε απαλλαγή. Αυτή πρέπει να παραμείνει η θέση μας και ακόμη και αν το Συμβούλιο δεχθεί το non-paper και το βάλει στην ημερήσια διάταξη του Κορεπέρα, ακόμη και τότε, και το είπα στην εισαγωγή μου, νομίζω ότι δεν μπορούμε να χορογήσουμε την απαλλαγή, διότι για αυτή την απαλλαγή δεν έχουμε τις πληροφορίες που ζητήσαμε. Αφού διαπιστώσαμε ότι δεν λαμβάναμε τις πληροφορίες, θελήσαμε να δημιουργήσουμε τις περιστάσεις που θα επιτρέψουν, νομίζω, στον διαδοχό μου που θα είναι υπεύθυνο για την απαλλαγή 2016 να εργαστεί σε ένα καλύτερο ε, κλίμα που όπου θα μπορεί να θέτει γραπτές ερωτήσεις για τις οποίες θα λαμβάνει απαντήσεις όπου θα υπάρχει μια πραγματική ανταλλαγή πληροφοριών όπως έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με όλα τα άλλα όργανα τα θεσμικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς όπου έχουμε ομαλές σχέσεις μαζί τους και δεν έχουμε ομαλές σχέσεις με το Συμβούλιο. Συμβούλιο. Το πλεονέκτημα τώρα είναι ότι η απαλλαγή θα ψηφιστεί τον, στο δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου. Έχουμε λοιπόν ακόμη λίγο χρόνο και αν μέχρι τότε βλέπουμε ότι τα πράγματα εξελίσσονται αρκετά ικανοποιητικά στο Συμβούλιο θα μπορούσαμε ακόμη να προσθέσουμε μια παράγραφο ε, στην εκθεσή μου για να γίνει πιο θετική. Αλλά να χορηγήσουμε την ε, απαλλαγή. Εγώ ως εισηγητής πρέπει να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι δεν είμαστε ε, τώρα σε θέση να το πράξουμε. Ευχαριστώ θερμά. Ολοκληρώσαμε και αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης και έτσι περνούμε στο σημείο 6 και καλώς ορίζω θερμά τον Επίτροπο Χάν, Επίτροπο Πολιτικής Γειτονίας. Πολιτική γειτονία, λοιπόν και πάνω απ' όλα οικονομικά της πολιτικής γειτονίας. Ας ε, αφήσουμε το χρόνο να μπουν και οι συνάδελφοι. Ο κύριος Τσέλερ είναι εδώ για το κεφάλαιο αυτό στον έλεγχο του προπολογισμού. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τις ευκαιρίες που είδαμε που είχαμε να αξιολογήσουμε την ε, βοήθεια που δίνεται στις χώρες γειτονίας, την Τουρκία, το Λίβανο, την Ιορδανία. Μιλήσαμε και με τους ε, πρέσβεις, οι οποίοι διαπιστώσαμε ότι πρέπει να δίνουν ε, ενημέρωση για την χρήση των κονδυλίων της πολιτικής γειτονίας. Έχετε το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Χάν. Συμφωνήσαμε με τους συνεργάτες μου να κάνω την παρουσίαση στα αγγλικά. Την έχω ετοιμάσει λοιπόν, είναι στα αγγλικά, μου την έχουν ετοιμάσει, είναι στα αγγλικά, για να μην χρειάζεται να την ξέρω ότι με μεταφράζω. Επιτρέψτε μου να σας την παρουσιάσω στα αγγλικά και μετά να κάνουμε τη συζήτηση και στα αγγλικά και στα γερμανικά αναλόγως. Ξεκινώ όμως ευχαριστώντας Πρώτον, γιατί ο πάγιο ενδιαφέρον. Δεύτερον, για την βούληση, ε, αντί να επαναπάβεστε στις δικές μας ε, αναφορές, να επισκέπτεστε και τις χώρες για να βλέπετε σώμα σε τη χρήση των κονδυλίων. Έχουμε εργαστεί μακρόν στα θέματα αυτά και είναι για μένα πολύ σημαντικό και με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να έχω αυτή την ανταλλαγή απόψεων για την πολιτική μας για να μπορώ και να δώσω τις πληροφορίες, την ενημέρωση για τις στοχεύσεις της πολιτικής μας και βέβαια για να ενημερώνω και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε μερικές φορές γιατί ο στόχος μας δεν είναι η σωστή αξιοποίηση των κονδυλίων, η χρηστή διαχείρισή τους, αλλά η αξιολόγηση του πόσο χρηστή, πόσο σωστή και αποτελεσματική ήταν η χρήση τους. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ στη συνομιλία μαζί σας. Και πέραν βέβαια της σημερινή συνάντηση. γιατί Θέλουμε πάρα πολλά να σας εξηγήσουμε ποιες είναι οι επιλογές μας και να εξετάσουμε από κοινού ε, ποιες, ποιοι είναι οι περιορισμοί στις δυνατότητες δράσεις. Μπορεί να μην έχουμε μπει ακόμη στον κύκλο της διαδικασίας απαλλαγής, αλλά θα ήθελα όσο το δυνατόν βέβαια σύντομα και με το βλέμμα και στο ρολόι να δώσω πολύ σύντομα κάποιες απαντήσεις σε θέματα απαλλαγής και γι' αυτό επιτρέψτε μου να περάσω για λόγους συντομίας στα αγγλικά για να δώσω και τις απαντήσεις όπως τις έχει στήσει Πρόεδρος και προχωρώ στα αγγλικά. Με δεδομένο λοιπόν το πλαίσιο αλλά και τις προτεραιότητες όπως τις έχουμε ορίσει στην πολιτική γειτονία για την περίοδο 2017-2020 γιατί όπως ξέρετε βρισκόμαστε σε μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση αυτή τη στιγμή. Ήρθα για να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων η οποία είναι πάντα χρήσιμη για μας καθώς προχωρούμε και στην υλοποίηση της πολιτικής μας. Ταυτόχρονα αποδεικνύει τη χρησιμότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων ως μέσον άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Έτσι λοιπόν, καταρχάς για το 2015 και την αξιολόγηση της χρήσης των κονδυλίων και βέβαια τις εκθέσεις των ε, δημοσιονομικών ελεγκτών. Για το 2015 έχει επικριθεί η Επιτροπή ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει στο μέγιστο τα ποσοστά, στα μέγιστα ποσοστά τα ε, ποσά. Αυτά ισχύαν για το 2015-2016. Τώρα έχουμε ένα υπόλοιπο ελάχιστο ε, που αφορά και τη διαχείριση σε σχέση με τις ωφελούμενες χώρες. Επίσης, οι ανεξάρτητοι δημοσιονομικοί έλεγχοι αποδεικνύουν ότι στο δικό μας τομέα είχαμε ποσοστό σφάλματος κάτω από το 1% το 2016, που είναι πολύ μικρότερο από το όριο του 2% όπως είχε οριστεί. Φαίνεται από τους ελέγχους και τις εκθέσεις αυτές ότι έχουμε μπει στο σωστό δρόμο. Το 2016-2017 δημοσιεύθηκαν 8 ε, δημοσιονομική έλεγχη και για, την, ε, ε, για τις επιδόσεις της παρεχόμενης βοήθειας σε χώρες ωφελούμενες, αλλά και στην αποδοτικότητα σε σχέση με το στόχο της αντιμετώπισης μετανάστευσης. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε πιο συγκεκριμένη στόχευση όταν οι λόγοι δαπάνης, οι της δαπάνης δημοσιεύονται και ακολουθούν τις συστάσεις, πράγμα το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει και στη δική μας προσπάθεια, ώστε η βοήθεια, η χορηγούμενη να παρέχεται κατά τρόπο αποτελεσματικό και χρηστό. Και επίσης θα ήθελα να σχολιάσω το τελευταίο ότι το ελεγκτικό συνέδριο με τις εκθέσεις του μας ενθαρρύνει ούτως επίν και έχει κάνει και, με την πλευρά, και από πλευρά του σημαντική πρόοδο, γιατί θυμάμαι εκθέσει δημοσιονομικού ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο που στηριζόταν σε αυτοψίε ή σε ε, επισκόπηση τη κατάστασης στις ε, ωφελούμενε χώρες ε, που ανέρχονταν σε δύο ή τρία χρόνια πριν και είχαν ως εκ τούτου περιορισμένο πεδίο. Ε, το είχαμε άλλωστε επισημάνει και γι' αυτό θα ήθελα να σημειώσω ότι και το ελεγκτικό συνέδριο φαίνεται να αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες που έχουμε και εμείς από πλευράς μας εκφράσει και να έχει αντιδράσει κατά τρόπο πολύ θετικό. Θα ήθελα επί, επί παραδείγματι να αναφερθώ στον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου για την, ε, την Ισία, την οποία παρεμπιπτόντως ε, επισκέφθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, όπου καταγράφει το ελεγκτικό συνέδριο ότι έχουν δαπανηθεί σωστά τα χρήματα, έχουν στοχεύσει στο στόχο της ε, διασφάλισης της δημοκρατικής μετάβασης και της δημοκρατίας στη χώρα. Βέβαια η Τινησία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για περαιτέρω μελέτη εσωτερική των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σχέση με τις χώρες αυτές, γιατί όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι θα πρέπει να υποστηρίζουμε την ε, ε, δημοκρατική πρόοδο, αλλά οι παλινδρομήσεις ε, στη χώρα δεν είναι πάντοτε ότι καλύτερο και δεν επιτρέπουν πάντοτε την ανάπτυξη, η υλοποίηση μάλλον των στόχων με βάση τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες που έχουμε. Στον έλεγχο αυτόν το Ελεκτικό Συνέδριο επίσης εντοπίζει μεθόδους εργασίας που θα μπορούσαν παραδείγματι να ενισχύσουν περισσότερο το, στόχευση της ε, παρεχόμενης από μας βοήθειας. Επιπλέον πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο με τους εταίρους για τη βελτίωση της χρήσης της βοήθειας. Βέβαια το Ελεκτικό Συνέδριο μερικές φορές διατυπώνει σε ευρύ όρου τα συστήματα τις συστάσεις του και τις προτάσεις του, στοχεύοντας σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και όχι σε μακροπρόθεσμη υλοποίηση της, των στόχων. Σε σχέση με τον έλεγχο δηλαδή της απόδοσης πρέπει να διερωτηθούμε αν υπάρχει κάποιο όριο. Δηλαδή αν κάπου χαράσουμε τη γραμμή από ποιο σημείο και μετά θεωρείται ότι έχει υλοποιηθεί ο στόχος. Φυσικά και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση του χρήματος του Ευρωπαίου Φορολογουμένου και να είμαστε αυστηροί στους ελέγχους, αλλά ταυτόχρονα όταν έχουμε να κάνουμε με αβεβαιότητα και αστάθεια σε πολλές από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμε θα... Ε, και που ασφαλώ έχετε και εσείς επισκεφθεί και το έχετε διαπιστώσει φαντάζομαι στις ε, αποστολέ σα. Έχουμε δύσκολες συνθήκες λοιπόν, οι οποίες θέτουν σε δοκιμασία ε, τις μεθόδους μας και τα διάφορα μέτρα. Αλλά το μεγαλύτερο σφάλμα θα ήταν να μην, συνεχίσουμε να προσπαθούμε ή να μείνουμε αδρανείς. Και εδώ πάλι το ζήτημα της μετανάστευσης θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως ένα εύστοχο παράδειγμα των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δρούμε, γιατί βεβαίω δεν είναι αποτελεσματικό το κάθε μέτρο που θα μπορούσαμε να φανταστούμε, αλλά καθώς έχουμε αντιμετωπίσει άνευ προηγουμένου, όχι ένα, αλλά πολλαπλά κύματα Μετανάστευση είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε. Και άπαξ και αντιδρά κανείς, βεβαίως κανείς δεν μπορεί να είναι αλάθητος, δεν μπορεί να είναι απαλλαγμένο από σφάλμα, άπαξ και υπάρχει δράση, μπορεί να υπάρξει και σφάλμα και στην εκ των υστέρων αξιολόγηση μπορεί να κριθεί ότι κάποιο μέτρο μπορεί να ήταν λιγότερο αποτελεσματικό από κάποιο άλλο, αλλά την ώρα που πρέπει να δράσουμε και να αντιδράσουμε και αυτό το λέω και για το μέλλον γιατί δυστυχώ βλέπω ότι θα παραμείνει στην επικαιρότητα το θέμα τη μετανάστευση. Αυτά που μάθαμε τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ασφαλώ θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για το ε, περαιτέρω δρόμο που έχουμε να χαράξουμε και τα μέτρα που θα υιοθετήσουμε για το μέλλον. Ε, γειτονία λοιπόν πολιτική διεύρυνση και προτεραιότητε στο δεύτερο ήμιση του τρεχοντος πολιτου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου 2017-2020. Δηλαδή η προσεχής ε, γενιά γειτονία είναι και είναι μάλλον και διεύρυνση ε, στοχεύει σε σταθεροποίηση, ορατότητα, ευελιξία και τέταρτον μεγαλύτερα αλλά λιγότερα ε, έργα, με μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας που θα έχουν τα μεγαλύτερα έργα, περισσότερη μόχλευση για τα όσα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερη ορατότητα, περισσότερη και καλύτερη επικοινωνία ως προς τα αποτελέσματα, επικοινωνία και επικοινωνιακή πολιτική. Η πολιτική γειτονία για το 2015 βλέπουμε να έχει μεταλλαγή σε μια διαφορετική προσέγγιση με ε, αποδοχή των προγραμμάτων για το 2016-2017 από πλευράς των αποδεκτών και βεβαίως ε, η σταθεροποίηση αλλά και η ενίσχυση ε, της στεναρότητας των εταίρων μας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ασφάλεια μετανάστευση. Εδώ προσφέρεται σταθεροποίηση βάσεως, βασική σταθεροποίηση αλλά και ευκαιρίες για τους πολίτες της περιοχής. Κεντρική προσέγγιση αυτή και προχωρώ στους γείτονες προς Ανατολάς με πολύ καλά αποτελέσματα. Στην διάσκεψη Ανατολικής Γειτονίας τον Νοέμβριο θα καταγραφούν η Ουκρανία και η Γεωργία, παραδείγματι, με σημαντικές ε, μεταρρυθμίσεις που ήδη αρχίζουν να δείχνουν πρώτα αποτελέσματα. Οι Ουκρανοί και οι Γεωργιανοί πολίτες μπορούν πλέον να υποφεληθούν της πλήρους αφελευθέρωση από την υποχρέωση του διαβατηρίου. Η συμφωνία σύνδεση με την Ουκρανία επίσης ξεκίνησε από τις αρχές του μήνα. Η οικονομική όρια, απασχολησιμότητα και κυρίως για τους νέους θα είναι κύριοι μοχλοί της συνεργασίας στην Ανατολική Γειτονία. Ε, ο τομέας βέβαια της ασφάλειας τόσο στην Ανατολική όσο και στην Νότια γειτονία δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Παρέχεται εκτεταμένη ε, υποστήριξη για την βελτίωση των συνθήκων της ασφάλειας στην ε, Μολδαβία, Ουκρανία, Λίβανο, Ιορδανία, την Ισία και για την περίοδο 2017-2020 έχουμε συμπεριλάβει και εκτεταμένη χρήση κοινών προγραμμάτων βοήθειας και πολιτικής επικοινωνιακής προκειμένου να ενισχυθεί και η ορατότητα της οικονομικής βοήθειας που προσφέρουμε στην πολιτική διεύρυνση με την προενταξιακή βοήθεια συνεχίζουμε την εστίαση στα βασικά καταρχάς με ε, αξιόπιστη, ε, αυστηρή αλλά και δίκαιη διαδικασία διεύρυνσης. Η προενταξιακή αυτή βοήθεια είναι ένα ε, αναντικατάστατο μέσο για την ικανοποίηση των βασικών προϋποθέσεων και όρων της διεύρυνσης και αυτό, σε αυτό το εργαλείο θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηριζόμαστε και για τα επόμενα χρόνια. Πρέπει όμως να δείξουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία αλλά και να επιδείξουμε μεγαλύτερη ορατότητα σχέση με τις χώρες και τις προοπτικές ενώ πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι θα ωφεληθούν από τη στενή ε, συνεργασία, ενοποίηση, προσέγγιση και οι πολίτε εν ώψη ε, διεύρυνσης ε, πρέπει να δούμε όλα τα στοιχεία και ασφαλώ αυτό θα σας ενδιαφέρει. Στην περίπτωση της Τουρκίας μας ανησυχεί ακόμη η κατάσταση στην Τουρκία και κυρίως η ε, κακές επιδόσεις σε σχέση με κέρια πολιτικά κριτήρια για τα οποία δεν μπορούμε να δείξουμε ε, αμέλεια. Η να επαναπαυόμαστε. Πρέπει να απαιτήσουμε από την Τουρκία να τηρήσει τους όρους ε, με αυστηρούς τόνους. Παραμένει βέβαια ανοιχτή η πόρτα του διαλόγου για οικονομικές ανταλλαγές. Πρέπει να στηριζόμαστε και στη συνεργασία για τη μετανάστευση. Αλλά αυτό δεν μπορεί να σημαίνει ότι θα αποστρέψουμε το βλέμμα από τα τεκτενόμενα στη χώρα, στο εσωτερικό της χώρας. Η προενταξιακή βοήθεια από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία δεν είναι εν λευκό επιταγή ε, στηρίζεται σε προϋποθέσεις, άρα πρέπει να σταματήσουν οι διώξεις στον χώρο της δικαιοσύνης. Έχουν καταστεί αντιπαραγωγικές ε, οι συνθήκες μετά το ε, πραξικόπημα ε, τομείς ε, της κοινωνίας των πολιτών, θεμελιωδών δικαιωμάτων, δραστηριοτήτες, εκπαιδευτικές, πανεπιστημιακές, πάνε, καλύπτονται ιδιαίτερα από το προενταξιακό ταμείο και κυρίως το ένα, και πρέπει να πω το 1 τρίτο του ήδη καλύπτει τέτοιου είδους δραστηριότητες. Κανονισμοί που έχουν να κάνουν με τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία προκύπτουν στις αρχές του 2018 και θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κατανομή των ποσών και την αποδέσμευση των ποσών. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή ήταν μια στομή επισκόπηση και προτεραιότητε για την πολιτική μα για τα επόμενα χρόνια. Περιμένω τι δικέ σα παρεμβάσει και με πολύ χαρά θα απαντήσω στι ερωτήσει σα. από τι οποίε ορισμένε ενδέχεται να έχουν πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο και έτσι θα σας παρακαλέσω να μου επιτρέψετε να σας απαντήσω και γραπτό σε αν χρειαστεί. Η κυρία Γκρέσλη, ευχαριστώ πολύ ε, παράληψή μου το ότι δεν χαιρέτησα την παρουσία εδώ εκπροσώπων του ελεκτικού συνεδρίου. Με συγχωρείτε και σας καλωσορίζω και πάλι. Κύριε Επίτροπε, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με την πολιτική γειτονία, κυρίως γιατί έχετε τόσα πολλά κράτη στα οποία έχετε να ενημερώ, για τα οποία έχετε να ενημερώσετε. Έχουμε την ετήσια έκθεση το Μάιο, τον Ιούνιο και με την ενημέρωση βέβαια που λάβαμε. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολη κατάσταση, αλλά ας μην χαθούμε στα επιμέρους ζητήματα, γιατί υπάρχουν θέματα που μας ενδιαφέρουν, πολύ συγκεκριμένα, και για τα οποία θέλουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Τέσσερις είναι συνάδελφοι. Στάσεις πρώτος. Ehm, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο για την ε, λεπτομερή του εισήγηση. Οι ερωτήσεις μου ίσως να είναι λίγο πιο πολιτικής φύσης ε, ε, γιατί μιλάμε για τη χρηστή οικονομική διαχείριση της πολιτικής γετνίασης και όλες τις ε, δραστηριότητες όπου έχουμε αφιερώσει ε, ενέργεια και χρήμα και θα ήθελα να εστιάσουμε την προσοχή σε ένα κομμάτι του κόσμου, της αντιπροσωπείας της οποίας είμαι εγώ μέλος, δηλαδή την αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ και την Κνέζετ. Πώς είναι δυνατή το να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ σε τακτά χρονικά, κατά τακτά χρονικά διαστήματα καταστρέφει τα project που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Λωρίδα της Γάζας και όχι μόνο project των κρατών ε, της Ένωσης αλλά και project των κρατών μελών. Για παράδειγμα υπήρχε ένα συγκεκριμένο project που είχε χρηματοδοτήσει, το, ε, χρηματοδοτήσει η χώρα μου το Βέλγιο και ε, ε επανειλημμένα Έχετε πει ότι, σας έχουμε πει και εμείς, ότι θέλουμε οι Ισραηλινοί να αποζημιώνουν τις καταστροφές αυτές σε έργα, οι project που έχει χρηματοδοτήσει η Ένωση. Πώς βλέπετε εσείς αυτήν, την, τη συνέχιση μάλλον αυτής της κατάστασης στο πλαίσιο της πολιτικής γετνίασης, γιατί και αυτό είναι ένα στοιχείο σημαντικό. Εμείς δαπανούμε εκατομμύρια για project τα οποία ε, ε, ε, καταστρέφονται. Είναι δηλαδή μια κατασπατάληση χρημάτων των φορολογουμένων. Επιπλέον εμείς ως βουλευτές δεν έχουμε καμία δυνατότητα πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας όπου ε, γίνονται και χρηματοδοτούνται διάφορα project. Υπάρχει όμως πρόβλημα ανεφοδιασμού σε ενέργεια και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία επενδύουμε κονδύλια τα οποία μετά δεν ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με θετικό τρόπο. Και το τελευταίο στοιχείο που με εκνευρίζει πολύ όταν το σκέφτομαι είναι το γεγονός ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανούμε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για ένα project που χρηματοδοτείται από τον ορίζοντα 2020 και δεν εμπίπτει άμεσα στη, ε, στους στόχους του ορίζοντα 2020 ένα project που λέγεται Low Train και αφο... Ε, το οποίο project λοιπόν δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Πολλοί νομικοί λένε ότι το project του έρχεται σε αντίθεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ξέρω πως δεν είναι της δικής σας αρμοδιότητας, αλλά από τη δική μας πλευρά ε, θα πρέπει, πιστεύουμε, να υπάρχει μια συνοχή. En naleving van de mensenrechten toch voor een aantal waarden. En, en, en mijn vraag aan u is, eh, hoe, hoe, hoe, hoe kan u daarin uh, een, een, een, een draai vinden om, om dat ten goede te keren?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 Äh, äh, ναι, ευχαριστώ πολύ. Πολύ επίκαιρη η ερώτηση. Και στο Ταλίν την προηγούμενη Παρασκευή με μια από τις συνεδριάσεις ε, του Γκίμλιχ ε, είχαμε την ευκαιρία να τη συστήσουμε. και να συστήσουμε μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών λοιπόν, εάν μπορεί να υπάρξει σχετική υποστήριξη για μια διεξοδική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορροφώνται και χρησιμοποιούνται κυρίως στην Παλαιστίνη. Κατά κεφαλήν η Παλαιστίνη λαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό ενίσχυσης από κράτος μέλους εκτός Ευρωπαϊκής, ε, ε, προς κράτος πέραν των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος κύριος και πρωτορχικός είναι η σταθεροποίηση της κατάστασης εκεί. Αλλά όχι η βελτίωση πολιτικά της κατάστασης. Απλώς ουσιαστικά είναι σαν να βάζουμε και να κρατάμε το καπάκι πάνω στον τέτζερι. Μέχρι στιγμής έχουν έρθει αποτελέσματα αυτά, αλλά δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση. Βέβαια και ενδέχεται να ενισχυθεί η πίεση και να μπορούμε πια να κρατήσουμε το καπάκι πάνω στο τέτζερι. Την επόμενη εβδομάδα στην Νέα Υόρκη θα έχω την ευκαιρία και πάλι να κάνω τις σχετικές συνομιλίες με το Γενικό ε, Διευθυντή, νομίζω τον λένε, της UNRWA, της ε, Οργάνωσης Λετωμένων Εθνών για την Παλαιστίνη και θα έχω την ευκαιρία να τον ρωτήσω εάν χρειάζεται επιπλέον κονδύλια πάλι ε, με όλο αυτό το δυναμικό, το δύσκολο που έχουμε, δηλαδή τα σχολεία που κλείνουν κτλ. Μια κατάσταση παράδεκτη για όλους μας και βεβαίως συμφωνήσαμε να κοιτάξουμε και ενώ ψη μιας λύσης των δύο κρατών πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα κονδύλια αυτά και με το σκοπό της εξυπηρέτησης των αναγκών σε ασφάλεια του Ισραήλ. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μόχλευση έναντι του Ισραήλ. Έχουμε μια προσέγγιση στη γειτονία σε μονοψήφιο αριθμό εκατομμυρίων για το Ισραήλ. Αλλά ταυτόχρονα λέμε ότι πρέπει να κοιτούμε ε, όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή αυτή, όχι μόνο δηλαδή την πολιτική γειτονία, αλλά να αναζητήσουμε κάθε δυνατό κορβανά που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Άρα θα μπορούσε στην απάντησή να δώσει άλλο συναδελφός ε, απαντήσεις. Αλλά ως θετική είδηση μπορώ να σας πω ότι η εύστοχη εδώ και χρόνια επίκριση του Κοινοβουλίου αλλά και άλλων για τα χρήματα σε ύψος εκατομμυρίων που διατίθεντο εδώ και χρόνια για υπαλλήλου στη Γάζα και δυσυνταξιούχους για τους οποίους δεν ξέραμε καν αν ε, μένουν εκεί εάν έχουν επαγγελματική δραστηριότητα ακόμη, εάν όχι. Ε, ήταν ένα θέμα λοιπόν το οποίο είχε δεχθεί πολλές επικρίσεις και αναλάβαμε την πρωτοβουλία από πέρσι και είπαμε ότι χωρίς να αλλάξουμε τίποτε στον όγκο των, ε, της παρεχόμενης βοήθειας είπαμε ότι για να ωφελήσει πραγματικά τη Γάζα αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο διατίθενται τα ποσά αυτά. Ιδάλλως είπαμε δεν μπορεί να είναι χρήσιμο αυτό. Και έτσι η Παλαιστινιακή Αρχή έκανε δεκτή αυτή την αλλαγή μεθόδου και αναπτύξαμε ένα σχέδιο σε ορίζοντα τριετίας έτσι ώστε πρώτα απ' όλα τα χρήματα αυτά να ενισχύουν μικρές μέσες επιχειρήσεις και να υπάρχει βέβαια και σχετική, ο έλεγχος. Δεύτερον, να προσφέρετε υποστήριξη σε οικογένειες που βρίσκονται σε ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια. αλλά και συγκεκριμένα ε, θελήσαμε να υποστηρίξουμε ένα έργο αφαλάτωσης υδάτων σε περιοχή η οποία κινδυνεύει να μην έχει πόσιμο νερό μέχρι το 2020. Ήταν λοιπόν οι πρωτοβουλίες μας τέτοιες, ώστε να καλύψουμε και τις ανάγκες σε χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Και βέβαια θα γίνει και η πολιτική αξιολόγηση τις επόμενες εβδομάδες. Η Πρόεδρος 7 έχω ακόμα στο κατάλογο. Παρακαλώ να είμαστε σύντομοι όλοι. Σταχόφσκι. Ευχαριστώ Πραγματικά πολύ μου άρεσαν αυτά που είπατε για το νερό που βράζει και το καπάκι και θα το χρησιμοποιώ και εγώ στις δικές μου ομιλίες γιατί πιστεύω πως εξηγεί πολύ καλά τι γίνεται στην ε, Ισραηλο-Παλαιστινιακή σύγκρουση και το πέταμα χρημάτων στην Παλαιστίνη. Ο συνάδελφος μιλούσε περισσότερο από την πυροπτική της Παλαιστίνης γιατί να χρηματοδοτεί η Ευρώπη ε, σχολεία από τα οποία έχουν το όνομα τρομοκρατών. Εγώ ωστόσο δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό, θέλω να μιλήσω για την Ισία. Πρόσφατα εδώ στην Επιτροπή μας διάβασα μια ανέκθεση του, Συμβουλίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με και νομίζω πως πολύ ωραία ε, συνοψίζει άλλες πληροφορίες ε, και εκθέσεις ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα για ένα σωρό project υπερβολικά πολλά τα οποία δεν έχουν παρά αποτελέσματα. Ε, όπως ας πούμε παράδειγμα έφερνε τα διάφορα project στην Ισία. Γι' αυτό και θέλω να πω, μήπως είναι καλύτερα να χρηματοδοτούμε ένα ή δύο project κλειδιά, να επιλέξουμε δηλαδή τα πιο σημαντικά όπως ας πούμε τη μεταρρύθμιση του διοικητικού μηχανισμού της χώρας, ε, η αποκέντρωση ή κάτι τέτοιο πάντως ε, σημαντικό που θα λύσει σημαντικά προβλήματα και θα φέρει τη χώρα πιο κοντά στο δρόμο προς τη δημοκρατία. Και πώς βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση στην ε, την Ισία. Θεωρείτε πως είναι ασφαλής και σταθερή η χώρα αυτή. Θεωρείτε ότι πρόκειται για μια χώρα που αρκούντος πληρεί αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Και έπειτα Μολδαβία. Ε, Εκεί πώς προχωράει η ε, έρευνα για τα κλεμμένα ευρωπαϊκά χρήματα και μετά φύρωμα. Κράτος που χρησιμοποιεί κάποιες φορές και το όνομα Μακεδονία και πραγματικά είναι σημαντικό να είχατε πει να βοηθήσουμε να σταθεροποιηθεί η χώρα. Ε, και προσέξαμε πολύ τα Βαλκάνια. Αλλά στο μέλλον τι θα γίνει, πώς θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει περαιτέρω την ΦΥΡΟΜ να σταθεροποιηθεί και να εκκριζώσει την διαφθορά από τη χώρα. Πώς θα εξασφαλίσουμε επίσης ότι εκεί θα επικρατήσει λιγότερη βία ή εν πάση περιπτώσει να μην τίνει προς κι άλλη σε συγκρούσεις και κοσυφοπαίδιο. Πώς βλέπετε την κατάσταση στο κοσυφοπαίδιο μετά από τις εκλογές, γιατί όταν δούμε ποιοι κέρδισαν σε αυτές τις εκλογές και ποιοι κατέχουν τώρα την εξουσία, Δεν ε, αναμένουμε να προχωρήσει πολύ γρήγορα η καταπολέμηση της διαφθοράς και τέλος Αλγερία. Η Αλγερία είναι ακόμα αξιοπιστή αφού Ναι, ναι, κλείνω, κλείνω. Αλλά σύντομα, κύριε Πίτροπε, είπατε ότι πρέπει να σας λούσουμε με τις ερωτήσεις μας και μετά θα επιλέξετε ποιες θα απαντήσετε και ποιες θα απαντήσετε γραπτός. Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω απάντηση σε όλα τα ζητήματα βέβαια. Την Ισία. Βεβαίω, η Ισία είναι ένα θέμα στο οποίο προσπαθούμε να αναπτύξουμε και να υλοποιήσουμε λιγότερα με έργα, αλλά μεγαλύτερα. Επίσης, είχαμε από πέρσι μια ανακοίνωση όπου αποφασίσαμε μέχρι το τέλος του 2020 να διπλασιάσουμε στα 300 εκατομμύρια ευρώ την ετήσια χορηγία προς την, την νησία με στόχο τη σταθεροποίηση. Και αυτό ήταν το θετικό. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είπα, μια συνάντηση για την εκπαίδευση κτλ. Είπαμε ότι θα ήταν τελευταία μέχρι τι επόμενε εκλογέ. Οι επόμενε εκλογέ είναι σε δύο χρόνια, θα δούμε. Υπάρχει περιπτώσει όμω, ε, υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τη σταθεροποίηση της οικονομίας πρέπει να κοιτάξουμε και ο τουρισμός βεβαίως τώρα έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων. Τώρα προσπαθεί να ανακάμψει. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η χώρα από τον τουρισμό, όπως άλλωστε και στην Αίγυπτο, όπου πρέπει να γίνει διαφοροποίηση στην οικονομία, διάφορα μέτρα έχουν σαν στόχο την ε, υποστήριξη της ενδοχώρας. Ξέρετε ότι στην ε, Τινησία υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πληθυσμού στις παράκτιες περιοχές. Στην ενδοχώρα είναι πιο αραιοκατοικημένες οι περιοχές, αλλά πρέπει να είναι στο ενδιαφέρον όλων μας να παραμείνει ο πληθυσμό αυτός εκεί που βρίσκεται, να μην αλλάξουν οι πληθυσμιακές ισορροπίες και άρα χρειάζεται και αυτή η υποστήριξη. Την τελευταία εβδομάδα υπέγραψα ένα επιπλέον πρόγραμμα 20 εκατομμυρίων ευρώ για ε, κέντρα πρωτοβάθμιας παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ε, ιατρικά κέντρα με ένα ε, επαρκές επίπεδο ποιότητας βέβαια, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του πληθυσμού στην ενδοχώρα. Προσπαθούμε λοιπόν να, είμαστε, να συγκεντρώνουμε τα έργα μας, αλλά ταυτόχρονα λόγω και των διαστάσεων αλλά και των μεγάλων αναγκών πρέπει να δραστηριοποιούμεθα σε διάφορους τομείς και μιλισμονούμε ότι την Ισία παραμένει αντιμέτωπη με σοβαρό πρόβλημα ε, ασφάλειας, τα σύνορα προς τη Λιβύη 600-700 χιλιόμετρα δεν με απατάει η μνήμη μου, ε, έχουν ανάγκη από φύλαξη και δεν είναι αμεληταίο αυτό. Ε, Μολδαβία. Νομίζω ότι από τόσο είπε ο Επίτροπος Ντόνκ είναι σαφής η κατάσταση γιατί είχε πει ότι εάν μπορεί να στοιχειοθετήσει τις δηλώσεις του, ας συνεχίσει, ας μας δώσει τις αποδείξεις. Εάν όχι, καλύτερα να μην μιλάει. Αυτό είχα πει, πέρασαν οι μέρες, πέρασε ο καιρός, δεν έδωσε καμία συνέχεια. Ε, δεν βλέπω δηλαδή να είναι βάσιμα τα όσα είπε. Κατά πάσα πιθανότητα αντιμετωπίζει προβλήματα απορρόφησης η χώρα. Και πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ των προβλεφθέντων ποσών και των ποσών ε, τα οποία πράγματι καταβάλλονται Αυτά θα καταβληθούν όταν πράγματι ε, προχωρούν τα έργα. Εάν δεν ε, κινηθούν αυτά τα χρήματα μπορεί να μην είναι σε θέση και να υλοποιηθούν τα προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι μπορώ, χωρίς να θεωρηθώ αφελής, να πω ότι είμαστε σε θέση να διαφοροποιήσουμε μεταξύ των όσων έχουν προβλεφθεί και των, των όσων έχουν σχεδιαστεί και των όσων υλοποιούνται. Οι κατηγορίες ε, ούτως ή άλλως από πλευράς του αναιρέθηκαν ύστερα από μια ανταλλαγή επιστολών ε, ούτως ή άλλως εγώ θα προτιμούσα να γίνει σχετική διόρθωση. Ε, ε, όπως και να έχει όμως ανερέθησαν αυτές οι κατηγορίες για την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έχουμε εν γέννη μια θετική εξέλιξη, όπως άλλωστε και στο Καουσφοπέδιο έχουμε μια ισχνότατη κοινοβουλευτική ε, πλειοψηφία με 61, 61 έδρας, έδρες έναντι 120 εδρών στο σύνολο του Κοινοβουλίου, πλειοψηφία 61 εδρών, ε, είναι προφανώς πάρα πολύ ισχνή αυτή η πλειοψηφία της μίας έδρας. Στο Κίμνιχ πάντως την προηγούμενη εβδομάδα μπορώ να σας ενημερώσω ότι είχαμε και με τον Υπουργό των Εξωτερικών το, της Βουλγαρίας αλλά και με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών ε, είχαμε την ευκαιρία να διαγνώσουμε βούληση για βήματα προόδου και τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη αντιλαμβάνονται τι έχει πάει στραβά τα τελευταία χρόνια και είναι διτεθειμένα να συμβάλλουν ώστε να μην υπάρξει παρεκτροπή η παρερμηνία της παρεχόμενης υποστήριξης. Κοσφοπέδιο. Έχουμε κυβέρνηση που μόλις έχει να καθήκοντα, είναι νωρίς ακόμη για να προβούμε σε οποιαδήποτε αξιολόγηση. Αλλού μπορεί να χρειάζονται τρει μήνε για να σχηματιστεί κυβέρνηση, εκεί χρειάστηκαν εννέα. Η σύνθεση ούτω ή άλλω τη κυβέρνηση δεν μπορεί να μας επιτρέψει μια σαφή ε, εικόνα ή προσδοκία για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πρέπει να περιμένουμε να αναλάβει δράση και σε σχέση με την αποδοχή από τους πολίτες. Η πρωτοβουλία πάντως του Προέδρου Βούσης για τον ιστορικό διάλογο στο Κοσμοπέδιο πρέπει να αξιολογηθεί θετικά, διότι πρόκειται για ένα μέτρο σημαντικό και που μπορεί να, να οδηγήσει και στην ανάπτυξη περαιτέρω βημάτων. Το Μαρόκο είναι πολύ σημαντικός εταίρος. Είμαι αισιόδοξο ότι οι ενοχλήσεις, ε, η δυσφορία η πρόσφατη σε σχέση με μια κρίση ως προς την αντιμετώπιση του θέματος της άδειας λειτουργίας κομμάτων Ε, σε σχέση και με την αποφάση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μπορεί να μπει πλέον ε, να θεωρηθεί ότι ανήκει στο παρελθόν. Η Αλγερία. Η Αλγερία έχει πάρα πολύ μεγάλο ποσό του πληθυσμού της στις παράκτιες περιοχές με τρόπο ζωής ε, που επηρεάζεται από τις υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου που για μας είναι άγνωστος. Έχει συνηθίσει ο πληθυσμός αυτός να έχει παγίως επιδότηση βασικών αγαθών. Οι παραδείγματα τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχουν δει καμία αλλαγή στην τιμή του καυσίμου τους. Ε, άρα υπάρχουν πολλά βασικά ζητήματα να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν. Εδώ και δύο χρόνια έχω ξεκινήσει με τις εσωτερικές οικονομικές ε, αρχές ή θεσμούς εντατική συνεργασία και αυτό βέβαια αφορά και άλλα κράτη, όχι μόνο, και, όχι μόνο την αλλεργία, αλλά πάντως μια στρατηγική συντονισμένη προσέγγιση για όλα αυτά τα κράτη τα οποία είναι σημαντικά για μας και σε θέματα που είναι σημαντικά για μας, όπως σε παραδείγματι την αποτελεσματικότητα στη χρήση τη ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ένα θέμα το οποίο βέβαια αφορά όχι μόνο την Αλγερία, αλλά και πολλές άλλες χώρες, ιδιαίτερα στα ανατολικά μας. Ευχαριστώ, Αγία Λαζέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Χάν που είστε για την εισήγησή σας και θα ήθελα να θέσω κάποιες ε, ερωτήσεις για την, Τινησία, την όπου ήμουν και εγώ την περασμένη εβδομάδα και εγώ την επισκέφθηκα. Πρέπει να συζητήσουμε όλα τα θέματα που αφορούν το Μαγρέμπ. Συμφωνώ μαζί σας απολύτως ότι το θέμα είναι να μετρήσουμε τους διάφορους κινδύνους προς τους οποίους εκτιθέμεθα όταν βοηθάμε κάποια χώρα. Και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και που είναι διατεθειμένοι να τους αντιμετωπίσουν. Όμως θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν ε, τρόποι ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτή τη χρηματοδότηση και να την ε, ε, στρέψουμε προς τη χρηματοδότηση του δημοκρατικού κόσμου της χώρας. Ε, μήπως θα μπορούσε δηλαδή να γίνει κάποιο, κάποια προσπάθεια ώστε το οικονομικό στρώμα που έχουμε με τις ε, ε, για να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες δίνει τη δυνατότητα στην Κομισιόν να μπει στα προγράμματα της χώρας και κατά πόσο θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με ένα δεύτερο επίπεδο βοήθειας. Βοηθάμε ναι μεν, αλλά όταν ερχόμαστε σε επαφή ε, θα πρέπει να απαιτήσουμε ότι ορισμένες από τις θεμελιώδεις κανόνες ε, για την ε, δημοκρατία ε, να επιμείνουμε να εφαρμόζονται. Ας πούμε, τέταρτη φορά να βλήθηκαν οι τοπικές εκλογές στην Τινησία, ε, πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν τελείως ε, ομαλά, ας πούμε, να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να συνδέσουμε αυτή την χρηματοδότηση με κάποια τέτοια ζητήματα, ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο να πούμε ναι μεν δηλαδή σας βοηθάμε, αλλά υπάρχει και μια προθεσμία, υπάρχει μάλλον ένα χρονοδιάγραμμα με κάποιες προθεσμίες, δεν μπορείτε να ε, παραλύετε το κράτος γιατί κινδυνεύουμε να έχουμε οπισθοδρόμηση όσον αφορά τους βασικούς κανόνες που θα έπρεπε να ισχύουν. Και θα μπορούσαμε δηλαδή έτσι να χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης ως μοχλό για να επιμείνουμε για κάποια τέτοια ε, ε, πράγματα. Ας πούμε και για κόσμο που μας ενδιαφέρει πολύ, για προκαθηγητές, για φοιτητές, ε, για διανοούμενους που θα μπορούσαν να δουν με διαφορετικό τρόπο τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιμείνουμε ώστε να μην ταπεινώνονται, να μην ταπεινώνονται γιατί πολλές φορέ, φορές ας πούμε δεν μπορούν να έχουν ε, θεωρήσεις για να έρθουν σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις. Να έχουμε δηλαδή ένα δεύτερο επίπεδο, σε αυτό το επίπεδο βοήθειας. Δεν είναι μόνο τα ευρώ που δαπανούμε ως βοήθεια ή τα, τα διάφορα project που κάνουμε ε, να είναι μια άλλη μορφή ε, βοήθειας και συνδρομής για την δημοκρατική σταθερότητα που μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Κάτι ακόμα για τις καλές πρακτικές. Και μιλώ για το Μαγκρέπ, δεν πάω στην Ουκρανία και θα λοιπά, γιατί μετά δεν θα σταματάω. Λοιπόν, να να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με πιο στεναρό τρόπο. Ας πούμε, μπορεί να είναι και η Μαυριτανία, μπορεί να... και η Κομισιόν το έχει αυτό να γνωρίσει. Κάναμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, ελπίζω πως θα είναι έτσι το αποτέλεσμα και στο τέλος να φτιάξουμε δηλαδή ένα σύστημα ιατρικής ασφάλειας, γιατί αυτό είπαμε και φέρνω και το παράδειγμα της Μαυριτανίας, ξέρω πως εσείς ε, εκεί δεν είστε αρμόδιος, αλλά στο Μαρόκο, στην Αλγερία, στην Τινησία θα μπορούσε να φτιαχτεί κάτι τέτοιο, ένα είδος ασφάλισης ιατρικής που θα προτείνουμε εκεί και που θα μπορούσε να έχει και αυτό μια λειτουργία. Και έπειτα άλλο η φάση θα μπορούσε να είναι πώς αυτές οι καλές πρακτικές θα λειτουργήσουν και πώς θα μπορέσουν να αποτελέσουν τμήμα αυτής της ε, στήριξης. Και τέλος ορατότητα. Πριν από λίγο καιρό ήρθαμε στο, πήγαμε στο Μαρόκο και συναντηθήκαμε ε, με εκπροσώπους σημαντικών, σημαντικών project που έχουν ως βάση την ε, στήριξη και Είδαμε και διαπιστώσαμε ότι οι ίδιες οι εταιρείε που λειτουργούν εκεί δεν έχουν ε, κάποιες φορές ιδέα ότι υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαμε λοιπόν από κοινού, όπως κάνουμε στην Ευρώπη, να μπορέσουμε και εκεί να συγχρηματοδοτήσουμε project. Ε, τη διακόπτη, διακόπτη η Πρόεδρος. Ευχαριστώ, κλείνει ομιλήτρια. Κύριε Επίτροπε, ναι. Νομίζω όμως ότι είναι τόσο καλό παράδειγμα αυτό που αναφέρατε γιατί τις από χρόνια σχεδόν ε, διαπραγματεύσεων ε, κατέληξαν σε ένα πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα το καλοκαίρι. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η προθέση πάντα υπάρχει, το σχέδιο πάντα υπάρχει, αλλά υπάρχει και η υλοποίηση. Υλοποίηση, υλοποίηση, υλοποίηση αυτό είναι, αυτή είναι η λέξη κλειδί. Όταν λοιπόν υπάρχουν διαρκείς ανασχηματισμοί ή τακτικοί ανασχηματισμοί, ε, δεν βοηθάνε για τη σταθερότητα του κράτους. Και προσπάθησα και με την επίσκεψή μου την προηγούμενη εβδομάδα να ελαχιστοποιήσω ή δυνατόν ε, τον κίνδυνο και να δείξω ότι και ιδιαίτερα για τον πρόεδρο της χώρας που έχει πολύ μεγάλο ρόλο και βέβαια στην ηλικία των 91 ετών έχει δεδομένο κύρος. Ήθελα λοιπόν να πω και για την αλλαγή του Υπουργείου των Εξωτερικών αλλά και γενικότερα ότι θελήσαμε μια σταθερότητα, ορίσαμε ε, ορόσημα Και πρέπει να πω ότι αυτό μου το έχει δάξει βέβαια και η εμπειρία μου όλα αυτά χρόνια, ότι αν είμαι σήμερα και μου πει κάποιο μέχρι το τέλο του 2019 το έχω κάνει, ε, δεν θα έχει υλοποιηθεί το 2019 εάν δεν έχουμε βάλει τριμηνιαίους στόχου, ορόσημα. Αυτό προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε και για το σε αυτό αναπτυξιακό πρόγραμμα, να ορίσουμε ορόσημα Ποιο θα πρέπει να έχει επιτύχει τι, και αυτό το είδαμε και με την Ελλάδα βεβαίω, ένα κατάλογο ο οποίος θα πρέπει να είναι δημόσιος, να δημοσιοποιείται ώστε να ασκείται και σχετική πίεση ώστε να μπορεί να παρακολουθεί και, οι να παρακολουθούν και οι πολίτες ότι πράγματι υλοποιήθηκαν τα ορόσημα ε, και βέβαια γι' αυτό μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά αισιόδοξο για τη χώρα αυτή. Δημοσιονομική υποστήριξη που αναφέρατε κι εσείς. Ε, νομίζω ότι αυτή η έννοια που χρησιμοποίησατε μπορεί να οδηγήσει και σε παρερμηνίες, διότι ε, υπενήσετε ότι προσφέρουμε χρήματα κατευθείαν στον ε, προϋπολογισμό της χώρας, της θυμησίας ε, κάτι το οποίο βεβαίως δεν είναι ε, στο σωστό και δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Όχι, εμείς έχουμε την υποστήριξη ε, προγραμμάτων στην αρχή και μέχρι το τέλος τους, που όμως μέσα από τον προϋπολογισμό θα χρηματοδοτηθούν. Επί παραδείγμα, τη μεταρρυθμίση χώρο της δικαιοσύνης θέλουμε να υποστηρίξουμε θα πρέπει να περάσουμε μέσα από τον προϋπολογισμό της χώρας και βέβαια εκεί και η μεταρρύθμιση των κρατικών δομών, των δημόσιων ε, δομών ε, πρέπει να προχωρήσουν. Όπως και το Εθνές Μαθηματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν ζητήσει, θα πρέπει να υπάρχει μια χρηστή δημοσιονομική διαχείριση από τις κρατικές αρχές, από τις δημόσιες αρχές, με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές για την Τινησία πάντα. Και βεβαίως ε, είπατε πολύ σωστά ότι η ορατότητα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το λέμε πάντοτε σε όλες τις συμφωνίες μας περιλαμβάνουμε αυτούς τους όρους. Και στην προηγούμενη μου θητεία ως Επίτροπος σε θέματα περιφερειακής πολιτικής είχα δει ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ε, σκέλος της αποτελεσματικότητας της πολιτικής μας, να υπάρχει ορατότητα, να μπορεί κανείς να βλέπει ότι ένα κτίριο έχει χρηματοδοτηθεί και βεβαίως ε, πιστεύω ότι θα έπρεπε ίσως ακόμη και να προσδιοριστεί σε ένα τεχνικό δελτίο που σε ποιο σημείο του πίνακα ε, του έργου θα πρέπει να αναγράφεται ότι συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι η χρηματοδότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι επαρκής η ορατότητα αλλά Πιστεύω επίσης, για να βελτιωθεί αυτή η ορατότητα, ότι υπάρχει και μια άλλη λύση, ότι σε κάθε ταμείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπάρχει ο όρο ΕΟΥ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε παραδείγματι το Ταμείο Μάντατ, που είναι το Ταμείο για την υποστήριξη τη χρηματοοικονομική πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Συρία. Ε, το λένε λοιπόν Ταμείο Μάντατ στα αραβικά μάλιστα έχει άλλο όνομα. Κανείς όμως δεν μπορεί μέσα από το όνομα αυτό να διαγνώσει ότι είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν εγώ είπα ότι πρέπει να ονομάζεται EU Syria Trust Fund, ε, καταπίστευμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Συρίας, το ίδιο και για την Αφρική. Να υπάρχουν μέσα οι όροι τα αρχικά Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μπορεί να είναι ένα ωραίο παιχνίδι να σχηματίζουμε ονόματα για τα ταμεία, αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κάτι το τετριμένο το ζήτημα της ορατότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάραντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω ε, δύο περιοχές στη γειτονία μας υπόψη μου και δύο σύντομες ερωτήσεις. Αναφέρατε πολύ σωστά ότι ότι είπα για την ε, Τουρκία ε, δεν θα έπρεπε να δίδεται η βοήθεια αυτή χωρίς όρους. Όταν ε, δίνει ένα πρόγραμμα 10 εκατομμυρίων στην Αίγυπτο για την ποινική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχουν όρις, διότι ο, ο πρόεδρος Σίση ίσως χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για διαφορετικό στόχο και σκοπό ε, για να στείλει ορισμένους αντιφρονούντες ε, στην φυλακή, παρόλο που είναι και μικρό το ποσό. Και δεύτερον, δεν συμφωνώ με τον Ντόναλτ Τραμπ, αλλά έχει ε, λάβει λογική απόφαση να κρατήσει 80 εκατομμύρια ε, ε, δολάρια από την βοήθεια στην Αίγυπτο λόγω ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Δυτική Σαχάρα τώρα, από ό,τι γνωρίζω, είναι η μόνη περιοχή όπου η Επιτροπή και ο Μηχανισμός Ευρωπαϊκής Γειτονίας και για αυτός για την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν υποστηρίζει την κοινωνία των πολιτών. Ξέρω ότι ε, χρησιμοποίησατε τη λέξη ανθεκτικότητα και η Σαχράουη ε, στην Αλγερία, στα καταβλισμούς των ε, μεταναστών νομίζω ότι αξίζουν αυτή την υποστήριξη διότι έχουν αποδείξει ότι ξέρουν πώς να οργανώνουν την κοινωνία των πολιτών. Και από την άλλη πλευρά και πάλι ε, μην σκεφτείτε ότι είναι κριτική, ε, διότι ξέρω ότι υπάρχει διαρθρωτική οργάνωση της Κομισιόν και ε, πώς κατανέμονται οι ευθύνες και τα χαρτοφυλάκια. Η Επιτροπή έχει αποφασίσει να δώσει κάποια βοήθεια για την ανάπτυξη στην Δυτική Σαχάρα της αλληλείας από το Μαρόκο. Και ξέρω ότι η Δυτική Σαχάρα είναι ε, ε, κατεχόμενη περιοχή από το Μαρόκο. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου και ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Ναι, τα 10 εκατομμύρια στην Αίγυπτο. δεν είναι κανένα ποσό για μένα με επιτέω. Και βεβαίως θα πρέπει να γίνει σωστά η διαχείριση και η διάθεσή τους. Τώρα, εάν πρόκειται για ένα ποσό του North African Window για την Αφρική σε συσχετισμό με ε, απαιτήσει που έχουν διατυπωθεί της Αιγύπτου για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, είναι δηλαδή ποσά τα οποία βοηθούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μετανάστευσης όπως αυτό προκύπτει σε επίπεδο Αιγύπτου. Πρέπει να πω ότι δεν γνωρίζω να έχουν διατεθεί ποσά άλλα πέραν αυτού παραδείγματι για το τομέα της δικαιοσύνης. Επίσης θα πρέπει να πω ότι για την πολιτική κοινωνία η Αίγυπτος είναι η σημαντικότερη για μας χώρα στην περιοχή αυτή. η Ουκρανία, η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι οι τρεις στρατηγικά σημαντικές χώρες στη γειτονία. Για λόγους κοινωνικο-δημογραφικούς και κοινωνικο-οικονομικούς μάλιστα, για μένα η Αίγυπτος είναι η μεγαλύτερη πηγή ενισχυών, γιατί έχει καθαρή αύξηση του πληθυσμού της κατά 7.000 ανθρώπους την ημέρα, 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα δεν μπορεί κανείς να ε, ε, δεν μπορεί να συγκρατήσει κανείς αυτή την εξέλιξη. Έχει πολλαπλασιαστεί ο πληθυσμός μας τα τελευταία έξι χρόνια, παραμένουν όμως πάντα στα ίδια γεωγραφικά όρια. Ξέρουμε ακόμα και από την εποχή τη βιβλική ότι είχε μεγάλη παραγωγή ε, σιτηρών η Αίγυπτος εξήγε ε, διαχρονικά σιτηρά, τώρα αναγκάζεται να εισάγει. Ταυτόχρονα γίνεται ε, σημείο διέλευσης μεταναστών σε μεγάλο βαθμό. Εάν όμως τα πράγματα ανατραπούν, θα μπορούσε να αποτελέξει ακόμα και πηγή μεταναστευτική. Και αυτό σημαίνει ανατροπή όλων των δεδομένων των σχετικών με τις μεταναστευτικές ροές όπως τις γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό πρέπει να συγκρατήσουμε αυτό το κίνδυνο Γι' αυτό και ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, βοηθήσουμε στην ε, σταθεροποίηση της χώρας, πάντοτε και με το βλέμμα στις δημοκρατικές εξελίξεις, αλλά ταυτόχρονα πρέπει και να ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στην ε, πράξη, να, να είμαστε και ρεαλιστές, τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί. Δυτική Σαχάρα. Έχουμε δύο διαφορετικά καταβλισμούς και διαφορετική αντίληψη σε σχέση με τους καταβλισμούς. Άλλη αντίληψη έχουν τα κράτη που είναι πολύ κοντά στο Μαρόκο Και έτσι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αρκετά ασαφή. Και εμείς που επηρεάζει βέβαια τι δυνατότητε να προγραμματίσουμε το μέλλον. Βεβαίως και όσο δεν έχει διευρυνθεί το θέμα αυτό και μέσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση εσωτερικά δηλαδή, δηλαδή, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και βέβαια το θέμα των αλλιέων είναι ένα ζήτημα που αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ευχαριστώ. κύριο Τσέλερ έχει το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τον Επίτροπο που ήρθε εδώ σε τόσο προχωρημένη ώρα. Αναφερθήκατε και στην εισαγωγική σας παρέμβαση στην απαλλαγή για το 2016. Έχουμε τα στοιχεία της Γενικής σας διεύθυνσης, ε, διεύθυνσης αλλά όχι την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου όταν έχουμε και αυτό στα χέρια μας νομίζω θα μπορούμε να κοιτάξουμε με ε, ακρίβεια τα στοιχεία της, της απαλλαγής του 2016 και να κάνουμε τη σχετική ανταλλαγή απόψεων. Μας είπατε ότι έχει πέσει κάτω από το επίπεδο του 2%, από το όριο του 2% το ποστό σφάλματος, χάρη στην καλή δουλειά των υπηρεσιών σας, αλλά και το ελεγκτικό συνέδριο πιστεύω έχει επιτοπλίστων στραφεί στην αξιολόγηση του εάν επιτεύχθησαν οι στόχοι που είχαν οριστεί με τα ποσά που δαπανήθηκαν ή αν απλώς ε, έκλεισαν κάποιες τρύπες ή ε, έγιναν ε, εμβαλωματικές παρεμβάσεις. Ο τομέας των αρμοδιοτήτων σας βεβαίως πιάνει από το, η περιοχή της Καυκασίας μέχρι το Μαρόκο και είναι πολλή δουλειά που έχετε αναλάβει συσύφιο έργο πολλές φορές. Έχουμε και τις έκτακτες εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου που κατά καιρούς έρχονται όπως παραδείγματι με το δημοσιονομικό έλεγχο για την Ουκρανία που δείχνει ότι υπάρχουν προσπάθειες, ότι γίνονται προσπάθειες αλλά όχι πάντοτε επιστεγασμένες με την επιτυχία που θα θέλαμε ή θα περιμέναμε από τις χώρες αυτές. Ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι και οι δικές μας επισκέψεις και παρεμβάσεις έχουν να κάνουν πάνω απ' όλα με τους πολίτες των χωρών αυτών. Το είπε και η Ίγκεμπορκ ότι θέλουμε και οι πολίτες να αντιλαμβάνονται τους στόχους των δικών μας επισκέψεων. Γιατί είναι όλο και πιο έντονη ανεπομονησία προς τις προσδοκίες για το τι μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση θυμίζω την αντίληψη των πολιτών της πρώην Ανατολικής Γερμανίας κατά την εποχή της ενοποίησης που λέγανε ε, εγώ πάω στο, στη Γερμανία, στη Δυτική Γερμανία, δεν έρχεται και το γερμανικό μάρκο σε μένα. Αντίστοιχα λοιπόν νομίζω ότι περιμένουν ανταπόκριση οι πολίτες των χωρών αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό πρέπει και να ενισχυθούν ε, οι δημόσιες αρχές υπηρεσίες, να υπάρξει οικοδόμηση του δυναμικού, αλλά ταυτόχρονα και να ενισχυθεί ε, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η εμπιστοσύνη στο τρόπο λειτουργία της δικαιοσύνης. Για την πολιτική γειτονία, πολιτική διεύρυνση ω καθήκον βέβαια ως αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, το ανέφερε και η Ίγκεμπορκ, κάνει το έργο της Επιτροπή, αλλά πρέπει και οι διπλωμάτε πρέσβεις και λοιποί να συμβάλλουν με, δική τους, ε, το δικό τους μερίδιο στην ε, ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Πιστεύετε ότι επιτελούν το μερίδιο που τους αναλογεί οι διπλωμάτες των κρατών μελών ή μήπως ε, κάποιοι προσπαθούν να αποκομίσουν κάποιο πολιτικό όφελος ίδιων ή υπάρχουν κάποιοι άλλοι συναγωνιζόμενοι ή ανταγωνιζόμενοι στην περιοχή αυτή Κίνα, Ρωσία, οι οποίοι μπορεί να ασκούν επιστολές πιέσεις προς τα Δυτικά Βαλκάνια ή και άλλες περιοχές του κόσμου και ταυτόχρονα να εκβιάζουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να εκβιάζουν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να λένε αφήστε τους αυτούς και ελάτε σε εμάς. και δεν θα έπρεπε να επιδιώξουμε σε όλα αυτά τα θέματα της γειτονίας να έχουμε μια απόλυτα συντονισμένη συνεργασία όλων των αρχών και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε ναι, το ξέρουμε ότι με το χρήμα δεν μπορούν να επιτευχθούν τα πάντα, αλλά με το χρήμα ε, υλοποιούνται κάποιες δομές οι οποίες μπορούν να στηρίξουν τα οικοδομήματα. Ευχαριστώ. Απάντηση. η αναφορά στο Σύσυφο για μένα σημαίνει την ερμηνεία που έδωσε στο μύθο ο Αλμπερ Καμιού και άρα μπορώ να πω ότι είμαι και ευτυχισμένος. Για όλα αυτά τα κράτη όμω, είτε πρόκειται για κράτη γειτονία, είτε πρόκειται για κράτη διεύρυνση, πρέπει να κοιτάξουμε σε ένα ορίζοντα πέστρων ετών το βαθμό πρόοδου και εκεί νομίζω θα αναγνωρίσουμε για τα περισσότερα κράτη πρόοδο. Εάν κοιτάμε την κατάσταση από τώρα ένα μήνα στον άλλον ή ακόμα και μέσα σε μια χρονιά, σε ένα δωδεκάμινο, ασφαλώς υπάρχουν εκλειδονισμοί, σκαμπανεβάσματα. Η Βοσνία Αρσεγοβίνη, επί παραδείγμα, το 2016 ήταν ένα κράτος το οποίο με πολύ μεγάλο θαυμασμό παρακολουθούσαμε όλοι γιατί είχε φοβερές πρόοδους. Ε, τώρα βλέπουμε ότι έχει συνθλιβεί από το βάρος των επιτυχιών της και προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της. Ένα καμπανέβασμα λοιπόν διαρκές, αλλά ταυτόχρονα και μακροπρόθεσμα μπορώ να πω ότι υπάρχουν σαφή αποτελέσματα, θετικά αποτελέσματα, που ίσως είναι δύσκολο να διαγνωστούν εάν κοιτάξει κανείς σε ένα στενό ορίζοντα ή μόνο πάνω σε ένα πρόγραμμα την επιτυχία να την κρίνει. Πρέπει να κοιτάξουμε όμως ένα ευρύτερο πεδίο, πρέπει να κοιτάξουμε την συνέχεια, την διατήρηση μιας συνοχής και συνέπειας στην υλοποίηση και γι' αυτό νομίζω ότι μπορώ να πω ότι για τα κράτη της Δυτικών Βαλκανίων και γενικά και της Ανατολικής Γειτονίας ιδιαίτερη έμφαση θα έδινα εγώ την ε, μετάβαση η μετατόπιση των προσπαθειών μας από το εθνικό στο περιφερειακό, στα περιφερειακά, ακόμα και τοπικά επίπεδα στην κάθε χώρα. Γιατί δεν λειτουργούν πάντοτε ε, η διάβλη επικοινωνίας, δεν, λειτουργεί, δεν λειτουργούν πάντοτε όσοι συγκοινωνούν τα δοχεία το εθνικό με τα περιφερειακά και τα τοπικά επίπεδα. Αυτό θα πρέπει να καλλιεργήσουμε περισσότερα. Εκεί θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας και βεβαίως αυτό συμπεριλαμβάνει και τις δικαστικές αρχές. Έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα αστυνομίας, ε, αστυνόμευσης που λειτουργεί και ως παρακαταθήκη του κομμουνιστικού καθεστώτος, αλλά αντίστοιχα το δικαστικό σύστημα δεν λειτουργεί και πρέπει να δημιουργηθεί ουσιαστικά Μην ξεχνάμε ότι για τη Δυτικά ε, Βαλκάνια δεν μιλούμε για διαδικασίε διεύρυνση, αλλά για μια, για μια ε, γενικότερη διαδικασία ε, όπου η βιωσιμότητα των προσπαθειών έχει πολύ μεγάλη σημασία με πρώτη και κυρίαρχη την καταπολέμηση της διαφθοράς Άρα πρέπει όχι μόνο όπου υπάρχουν προβλήματα να καταγγέλλονται και να διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και το επόμενο βήμα, δηλαδή της παραπομπής στη δικαιοσύνη και της κρίσης από τη δικαιοσύνη. Ε, και βεβαίως να μην περιοριζόμαστε στο φαινόμενο που σε πολλές χώρες καταγράφεται της δίωξη βάρος του μικρού ψαριού, όπως τα λέγαμε, και της... Ε, ε, ανενόχλητης δράσης των μεγάλων, ε, των μεγάλων καρχαριών, αλλά θα πρέπει όλοι να βρίσκονται ισότιμοι απέναντι στον ε, νόμο. Στα Βαλκάνια, πάντως στα Βαλκάνια, έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων για αυτή την ε, περίοδο, πολύ ψηλά. Και εκροή πληθυσμού, αναγκαστικά κάτι το οποίο έχουμε γνωρίσει και στις δικές μας χώρες στο παρελθόν. Και θα πρέπει να σημειώσω εδώ το γεγονός και μόνο ότι ξεκινήσαμε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ε, Σερβία οδήγησε σε μια πολύ σημαντική αύξηση των εξωτερικών επενδύσεων και μάλιστα όχι μόνο από τις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, από ευρω... επιχειρήσεις των ε, κρατών μελών δηλαδή, αλλά από διεθνείς επενδυτές και αυτό σημαίνει ότι ενισχύθηκε η αίσθηση εμπιστοσύνης στην ε, επικράτηση του κράτους δικαίου, στην κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα αυτή, με τις επενδύσεις που οδήγησαν σε θέσεις εργασίας, που οδήγησαν σε μείωση της ενεργείας και άρα των αριθμών των νέων που έφευγαν στο εξωτερικό. Ε, και αυτό το βλέπουμε νομίζω και στα νεότερα κράτη-μέλη, αλλά και στα υποψήφια και πρέπει να το υπογραμμίσω, η συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες, υπεραδείγματι και πρέπει να το τονίσω αυτό, έχει πολύ κακή εικόνα παρουσιάζει, με απογοητεύει ιδιαίτερα και πρέπει να πω ότι με ενισχύει βαθύτατα. Αυτό ισχύει όπως είπα για τα κράτη της Βαλκανική, αλλά και τα νεότερα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, τα νεότερα κράτη-μέλη. Ε, αυτοί δηλαδή οι οποίοι για δεκαετίες δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχή στις εκλογές περίμενα εγώ ότι θα έσπευδαν στην κάλπη με την πρώτη ευκαιρία αλλά... Ε, αυτό δεν ε, συμβαίνει, δεν συνέβη και σε αυτό αισθάνομαι πολύ ε, απογοητευμένος. Πρέπει σε αυτό λοιπόν να κάνουμε προσπάθειες, στο να πείσουμε τον πολίτη να πηγαίνει στην κάλπη. Και επίσης και στην περιοχή γενικότερα, αλλά και σε σχέση με τους δικούς μας πολίτες. η αποδοχή σε πολιτικό επίπεδο ε, διαρκώς επανέρχεται και πρέπει να επαναλαμβάνουμε και να τονίζουμε διαρκώς ότι υπάρχει ότι παραμένει η προοπτική της ε, ένταξης για τις χώρες αυτές. Κοιτώντας όμως ε, στο ιστορικό των δικών μας κρατών μελών, δεν βλέπω πουθενά σε κανένα κράτος να διαγράφεται πλειοψηφία ή αποδοχή της ιδέας για την, αποδοχή, για εισαγωγή ένταξη στο και ενός κράτους μέλους και πρέπει να δούμε σε σχέση με τα Σκόπια παραδείγματι η μέθοδος του καρότου αλλά ταυτόχρονα και του ραβδιού μπορεί να είναι χρήσιμη μόνο εάν το καρότο τελικά μπορεί να του το δώσουμε του υποψηφίου να το φάει όταν έχει κάνει τη δουλειά που έπρεπε γιατί διαφορετικά αισθάνεται μεγάλη ε, απογοήτευση και, αίσθημα, και συνέστημα ματέωσης. Άρα λοιπόν πρέπει να προχωρούμε στην ενθάρρυνση και στην ανταμοιβή. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να εξηγήσουμε και στους δικούς μας πολίτες γιατί είναι σημαντικό να έχουμε μια Ευρώπη των 27-28 μέλων σταθερότητα, προοπτικές και ε, αποφυγή ενδοευρωπαϊκής ε, ανεπιθύμητης ε, ενδοευρωπαϊκής μετανάστευσης. Αυτά πρέπει να τα εξηγήσουμε. Και επίσης δεν μπορούμε να δεχθούμε εμείς οι Ευρωπαίοι, το λέω αυτό για να ολοκληρώσω, ε, να επιτρέψουμε σε κανένα να μας εκβιάζει. Είμαστε και με διαφορά η πιο ελκυστική αγορά στον κόσμο. Για τις χώρες αυτές είμαστε ο σημαντικότερος χρηματοοικονομικός και οικονομικός εταίρος και εμπορικός εταίρος 75% ε, του ε, εξωτερικού εμπορίου των κρατών της Δυτικής Βαλκανικής ε, αφορά χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάτι ακόμη το οποίο είδα στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια με την ολοκλήρωση ενός εσωτερικού οικονομικού χώρου στα Δυτικά Βαλκάνια είδαμε τα τελευταία δέκα χρόνια την ενίσχυση του εμπορίου των κρατών της Δυτικής Βαλκανική σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση να διπλασιάζεται και φτάσει 46 δισεκατομμύρια. Ενώ μεταξύ αυτό σε σχέση με, την, ε, με το εξωτερικό εμπόριο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των κρατών μελών παρέμειναν οι εμπορικοί όγκοι ε, ίση, δεν, δεν ενισχύθηκαν. Άρα λοιπόν χρειάζεται, όπως είπα, να πούμε ότι δεν λύνει κάθε πρόβλημα το χρήμα, αλλά ταυτόχρονα με τα χρήματα μπορούμε να έχουμε ένα μέσο μόχλευσης ε, και να βοηθήσουμε στις περιοχές αυτές την ε, παρουσία και την δραστηριοποίηση εκείνων των ελίτ που θα βοηθήσουν στην βελτίωση των όρων για τους πολίτες των κρατών αυτών. Σε αυτό πρέπει να, τα ενισχύσουμε τα κράτη αυτά για να διατηρήσουν την αηφορία, τη βιωσιμότητα καλύτερα των πολιτικών τους. Ευχαριστώ. Κύριος Λιμπεράτσικη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητέ ε, Επίτροπε, η, η ερώτησή μου είναι κάπως διαφορετική. Μάρτιος 2019. Ε, Δεν θα έχουμε πια την Ηνωμένο Βασίλειο στην Ένωση και βεβαίως θα έχουμε ένα έλλειμμα οικονομικό και εξετάζουμε περικοπές. Θα μπορούσατε να υποβάλλετε ένα τέτοιο πρόγραμμα περικοπών για την πολιτική γειτονίας. Δεύτερον, εάν βάσει των αποδόσεων, των επιδόσεων βλέπετε ε, τι διασπάθηση χρήματος γίνεται, εκεί μπορεί να γίνει περικοπή. Ε, και να δούμε ε, ποια χρήματα είναι παραγωγικά και ποια χρήματα δεν είναι παραγωγικά. Μπορούμε να περιμένουμε μια τέτοια εξέλιξη. Ευχαριστώ. Ναι, όπως πάντοτε, στην αρχή υπάρχει μια συζήτηση για το μέλλον. Αλλά είπα ότι θα υπερασπιστώ την πολιτική μας, όχι επειδή είμαι ο επίτροπος για αυτόν τον τομέα και επειδή αισθάνομαι υποχρεωμένος να το πράξω, αλλά είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να παρέχουμε τα μέσα για να συνεχιστεί αυτό το οποίο έχουμε αρχίσει. Έχω μια θεώρηση, ένα όραμα να υπάρξει μια ζώνη γύρω από την Ευρώπη, διότι ε, σήμερα έχουμε ε, βλέπουμε ε, πώς διαμορφώνεται η όλη κατάσταση, βλέπουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο περίγυρος. Βλέπουμε ότι σήμερα έχει αλλάξει το θέμα ακόμα και για την Ουκρανία. και αυτό δεν είναι κάτι διατηρήσιμο, δεν είναι κάτι βιώσιμο, κάτι αποδεκτό, διότι αυτό ασκεί πίεση πάνω μας και αυτό βεβαίως και για τον Νότο ισχύει. Πρέπει να δίνουμε τα κατάλληλα κονδύλια. Σήμερα έχουμε 20-25 εκατομμύρια μετανάστες πρόσφυγες στην Ευρώπη. ακόμα και εκτοπισμένοι, μετατοπισμένοι. Τόσα εκατομμύρια που στην χειρότερη περίπτωση προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπρεπε λοιπόν να παρέχουμε τα κονδύλια για αυτούς και ε, για να έχουμε μια καλύτερη κατάσταση χρειαζόμαστε να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές, να έχουμε έναν καλύτερο προϋπολογισμό, πώς να το ονομάσω, δεν νομίζω ότι όλη την εξωτερική δράση, τον προϋπολογισμό εξωτερικής δράσης πρέπει να μπει σε ένα καλάθι. Διότι τότε θα είναι ανάμεσα στην Ουκρανία και στο Κονγκό. Όλα μαζί. Πρέπει να έχουμε χρηστή οικονομική διαχείριση και πρέπει να κάνουμε διακρίσεις ανάμεσα σε διάφορα καθήκοντα ε, που πρέπει να είναι ο στόχος μας για να υπάρξει σταθερότητα. Βεβαίως, δεν ξέρω, η πρόταση της Κομισιόν σήμερα, βεβαίως το γεγονό ότι, μας, ότι έχουμε, θα έχουμε πρόβλημα προϋπολογισμού όταν με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι η συνεισφορά είναι μεγάλη του Ηνωμένου Βασιλείου και πρέπει να αντισταθμιστεί. Χρειαζόμαστε όμως ε, κονδύλια για τους στόχους αυτούς. Και αν εξετάστε ε, τα τα απρόβλεπτα γεγονότα τα τελευταία έτη, ήταν κυρίως ε, στις γειτονικές χώρες. Έχουμε την κρίση των προσφύγων, έχουμε τη Λιβύη, έχουμε την Ουκρανία και νομίζω ότι στις περιπτώσεις, περιπτώσεις μπορούμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση αλλά με πολύ χρηματοοικονομική βοήθεια. Προτάθηκε να γίνει κάτι παρόμοιο με τη Λιβύη, όπως με την Τουρκία. Υπάρχουν δύο δυνατότητες ε, δεν ξέρω, να τυπωθεί χρήματα από, τις, ε, από τα κράτη-μέλη. Σήμερα δεν βλέπω χρήματα στον προϋπολογισμό. Δεν είναι ε, δυνατόν να λαμβάνουμε συνέχεια αιτήματα χρηματοδότησης. Μι, μιλήσατε για τα δύο καταπιστευματικά ταμεία. Έχουμε λάβει 24 εκατομμύρια σε χρήματα από τα κράτη-μέλη και για την ε, Συρία 93. Όλοι μου λένε ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά ε, βεβαίως ε, είναι διαφορετική η κατάσταση επιτόπου. Βεβαίως βασίζομαι σε εσά ότι θα μας υποστηρίξετε, θα με υποστηρίξετε σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι το πρόβλημα. Είναι δυστυχώς τα κράτη-μέλη που προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα. Και αυτό δεν είναι πάντοτε προς το συμφέρον όλων μας. Αλλά είναι ένα θέμα πάρα πολύ περίπλοκο, το οποίο χρειάζεται μεγάλη συζήτηση. Η κυρία Σμιτ. Ευχαριστώ, Επίτρεπε, για τη συναρπαστική ε, συζήτηση και το χρόνο που μας αφιερώνεις. Και ήθελα να κάνω μια κάπως προκλητική ερώτηση συνολικά χρήματα υπάρχουν, ε, προ... βλέπονται προϋποθέσεις, σε ποιο βαθμό τηρούνται οι προϋποθέσεις. Ακούσαμε την ερώτηση για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Άλλωστε επισκεφθήκαμε και την περιοχή και είδαμε ότι έχουμε καταπλησμό Παλαιστινίων προσφύγων με ηλικία ανά των 60 ετών. Υπάρχει εδώ και 60 χρόνια αυτός ο καταβλισμός και μάλλον θα συνεχίσει να υπάρχει για τα επόμενα για τις επόμενες δεκαετίες και θα συνεχίσει να υπάρχει και θα τον χρηματοδοτούμε εμείς. Και όπως είπες, λέει ο Μιλήτρια και εσύ, ε, για την ΟΝΡΑ, ε, την ε, Οργάνωση των Εθνών για τους Παλαιστίνιους, που κάνει πολύ καλή δουλειά, νεαρούς, νεαρές, βοηθάει να τελειώσουν και τα σχολεία τους και μετά να πάνε και στο πανεπιστήμιο. Και όντω κάποιοι μπορεί να φτάνουν μέχρι το πανεπιστήμιο, αλλά μετά από αυτό 2% μόνο από τους νέους και κυρίω κυρίως για τα κορίτσια από τις νέες Παλαιστίνιες ε, μπορούν να προχωρήσουν στην απασχόληση, γιατί περισσότερε από αυτέ παντρεύονται και πια κάθονται σπίτι και ασχολούνται με τα παιδιά του. Και άρα πάνε χαμένα τα χρήματα αυτά. Τι πρέπει δηλαδή να κάνουμε και από ποιο σημείο μπορούμε ή πόσο καιρό μπορούμε να περιμένουμε να, ε, για να δούμε αποτελέσματα ή σε ποιο χρονικό όριο ή σε ποιο ε, ουσιαστικό όριο θα ορίσουμε, θα βάλουμε την αξιολόγηση της πρόοδου. Για δε την Τουρκία, εγώ θα ρωτήσω το εξή. Πόσο ακόμα θα ανεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο θα αντέξουμε ακόμα. Είπατε ότι υπάρχουν χρήματα τα οποία χορηγούνται με βάση τις προϋποθέσεις, τους όρους, ότι καταγράφονται πρόοδοι σε ορισμένα τομείς. Αλλά σε άλλους τομείς παραμένει το ερώτημα πόσο ακόμα θα ανεχθούμε αυτά που γίνονται, παραβιάσεις των δικαιωμάτων και το καθεξής. Και αυτά τα μέτρα και σταθμά, ποιος τα ορίζει, ποιος τα εφαρμόζει και ποιος ελέγχει την εφαρμογή τους. Βλέπουμε πολύ συχνά δηλαδή ότι μας παρουσιάζονται συνήθως τα καλά ε, έργα στις επισκέψεις μας, αυτά που έφεραν καλά αποτελέσματα, που υλοποιήθηκαν πλήρως κτλ. κτλ ενώ τα, αυτά που δεν τα έχουν πάει τόσο καλά ω έργα δεν μας παρουσιάζεται καν, δεν έχουμε την ευκαιρία καν να τα δούμε. Έτσι λοιπόν για να συνοψίσω πώς κρίνουμε την ε, επιτυχία των προγραμμάτων και μέχρι πού ανεχόμαστε, πόσα ανεχόμαστε σε σχέση με αυτά τα οποία θέλουμε να επαληθεύσουμε. Κύριος Τσέλερ, αν μου επιτρέπετε και εγώ θα ήθελα να συνεχίσω σε αυτό το, πνεύμα. Το εύρος των παρεχόμενων κονδυλίων είναι ένα ζήτημα, το άλλο όμως είναι και το, η δημοσιονομική διακήρυξη. Έχουμε μια πληθώρα προγραμμάτων στρατηγικών, ε, ιδεών κτλ. Τα οποία, εάν τα κοιτάξουμε και πιο αναλυτικά για να δούμε το ποσοστό της απορρόφησης, συχνά δεν είναι αυτό εύκολα διαγνώσιμο. Και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε να έχουμε πιο καλή επισκόπηση των πραγματικά διαθέσιμων ποσών διαθέσιμων για τους στόχους οποίους έχουμε ορίσει. Τι διάγνωση επίσης του πόσο, σε ποιο βαθμό υλοποιούν τους στόχους αυτούς αυτά τα κονδύλια και βεβαίως θα πρέπει με κάποιο τρόπο μέσα στα δύο-τρία χρόνια να είμαστε σε θέση να κρίνουμε εάν δεν έφεραν τα προγράμματα αυτά τα ορισθέντα ε, οριστέντα και αναμενόμενα αποτελέσματα. Πήγαμε στην Ιορδανία, ήμουνα και εγώ εκεί και με ιδιαίτερη έμφαση θέλω να εξάρω την ορατότητα και τη σημασία της ορατότητας των έργων που έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι 70% για την UNRWA, ε, UNRWA για τους ε, Παλαιστινίους, που όμως τελικά αναφέρονται στην εντολή τους ε, στα Ηνωμένα Έθνη και άρα δεν έχουν να μας δώσουν και λογαριασμό. Και επίσης είχα την ευκαιρία να συζητήσω με έναν ε, Παλαιστίνιο της, του Λιβάνου, ε, ταξιτζή στο Βερολίνο, αυτές τις μέρες που επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό που είπε η συνάδελφος ότι δηλαδή πληρώνουμε για τα σχολεία των νεαρών ε, Παλαιστινίων που μπορεί να πάνε και μέχρι το Πανεπιστήμιο, αλλά τελικά και το κράτος του ίδιου του Λιβάνου δεν τους επιτρέπει να ασκήσουν το επάγγελμα για το οποίο έχουν σπουδάσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει νομίζω να επιμείνουμε όλο και περισσότερο ε, να αλλάξουν πολιτική κράτη τα οποία είχαν ε, σε τελευταία ανάλυση μεγάλο όφελος από τα κονδύλα τα οποία εμείς διαθέτουμε. Ναι, ήταν ε, αρκετά, αρκετά εκτενής η παρεπίπτουσα παρέμβασή σου, αλλά εν πάση δίνω το λόγο στον Επίτροπο. Ναι, να σας πω. έχουμε αναλάβει ένα χαρτοφυλάκι, έχουμε αναλάβει ένα καθήκον και δεν έχουμε την πολυτέλεια να πάψουμε τη συνεργασία με τα κράτη αυτά, τα κράτη εταίρους, τα κράτη της γειτονία. για τελικά καθήκον μας είναι να συμβάλλουμε στην μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση της κατάστασης και κατά κανόνα αυτό είναι κάτι το οποίο κάνουμε σε συνεργασία με τις χώρες αυτές από κοινού. Θα σας δώσω και ένα παράδειγμα για να σας εξηγήσω αυτό που είπα ότι ένα-δύο χρόνια μπορεί να μην φτάνουν για να προβούμε σε μια αξιολόγηση της κατάστασης στον ε, χώρο των αραβικών κρατών. Και αυτό είναι βέβαια ζήτημα και παραδόσεων και νοοτροπίας. Επισημαίνεται σημαντικό έλλειμμα σε ανθρώπους με επαγγελματική και κατάρτιση, το vocational training που λέμε. Έχουμε ανθρώπους που έχουν πρακτική ε, γνώση ενός επαγγέλματος τεχνικού. Λοιπόν, διαθέτουμε εμείς ε, μέσα, τεχνικά μέσα, προγράμματα, υλικό, αλλά θα πρέπει να αλλάξει κοινοτροπία. για να μπορέσει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι έχει οικονομική αξία ε, και η ε, χειρονακτική δραστηριότητα. Για να μην πω ότι στις δικές μας χώρες ένας καλός τεχνίτης σε μεγάλο ποσοστό μπορεί να κερδίζει περισσότερα από ότι ένας ε, με πανεπιστημιακό πτυχίο. Άρα λοιπόν πρέπει και στις χώρες αυτές να δώσουμε αυτήν την ε, αλλαγή αντίληψης, να βοηθήσουμε στην αλλαγή αντίληψης και στην υλοποίηση και βεβαίως είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε. Θα πρέπει ταυτόχρονα να προτιμήσουμε ένα επιχειρησιακό ε, πεδίο, τοπίο, το οποίο θα διευκολύνει την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασία. Ε, προσπάθησα για τη Γάζα να συμβάλλω με την διάθεση των κονδυλίων που έχουμε να προσφέρουμε στην ε, ανάπτυξη νεοφιών επιχειρήσεων που θα οδηγήσουν και σε δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Ε, αλλά η Γάζα με 2 εκατομμύρια κατοίκων δεν μπορεί να χρειαστεί, δεν χρειάζεται 30.000 εργαζομένους, γιατί είναι σε τόσο κακή οικονομική κατάσταση η βάση οικονομική, γιατί είναι κατεστραμμένο τοπίο και άρα πρέπει να βρεθεί λύση και με το Ισραήλ ώστε να μπορούν να εισάγονται και να εξάγονται προϊόντα από τη Γάζα, προϊόντα της Γάζας να εξάγονται. Ωστόσο το Ισραήλ έχει επιβάλει περιορισμούς ως προς το εμπόριο. ως προς τον όγκο των εισαγωμένων και εξαγωμένων αγαθών και για λόγους ανησυχιών για την ασφάλεια. Και εδώ βλέπουμε ότι κλειδώνει το ένα πρόβλημα το άλλο και δεν είναι εύκολο να λύσουμε τα προβλήματα, αλλά καθήκον μας είναι να επιδιώξουμε να δώσουμε λύση στα προβλήματα. Η πολιτική των επικισμών, είναι παραδείγματι, δεν βοηθάει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας στη δυτική ε, ε, όχθη και δι των νεαρών Αράβων, του Ναντίον μάλιστα. Και βλέπουμε στους θύλακες καταρρεμημένο τον κόσμο αυτόν, όπου υπάρχει δυνατότητα για κάποια οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να συνδέεται με το εμπόριο κυρίως. Και άρα και εδώ θα πρέπει να αναζητηθούν και να δοθούν και πολιτικές λύσεις, χωρίς τις οποίες δεν μπορούμε να βγούμε από το αδιέξοδο, αλλά το θέμα είναι τι είδους ε, μέσω μόχλευσης ή πόσο ισχυρή μόχλευση μπορούμε να έχουμε ε, όλοι εμείς. Δεδομένου ότι δεν έχουν και 100% σύμφωνη αξιολόγηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην αναφερθώ στη νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί έχω επισκεφθεί πολλές φορές την ε, περιοχή και βλέπω πολλά πράγματα που δεν έχουν προχωρήσει και δεν έχουν ολοποιηθεί. Είναι πολύ περίπλοκα λοιπόν τα ζητήματα και δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα εξαντλήσουμε στη δημοσιονομική διαχείριση. Εμείς μπορούμε να έχουμε όλοι πολύ συγκεκριμένε ε, ε στοχεύσεις. Αλλά, και χωρίς να θέλω να πετάξω την μπάλα στην ε, εξέδρα, ε, θα σας απαντήσω στα σχόλιά σας ότι πρέπει να τηρούνται βεβαίως κάποιες προϋποθέσεις, οδηγίες, όροι κτλ αλλά και επειδή δεν μπορούν αυτοί οι όροι και οι οδηγίε να τηρηθούν, δεν μπορούν να αποδεσμευθούν τα κονδύλια. Έτσι αυτή είναι η αρχή. Ανάμεσα στην ιδέα και την ορίμανση ενό έργου, για την ευρωπαϊκή τουλάχιστον θεώρηση, έχουμε τεράστια απόσταση και απόκληση. Και αυτό είναι το πιο ε, δύσκολο πρόβλημα. Ακόμη και να πάμε να πούμε ότι κάνουμε απευθεία υλοποίηση. Ε, τελικά ε, τα πάντα θα κρυθούν από τη βιωσιμότητα των εγχειρημάτων και των έργων που θα αναπτύξουμε. Δεν μπορώ να πάω εγώ δηλαδή να κατασταθώ εκεί και να διοικώ την επιχείρηση που θα έχω στήσει, ακόμα και αν τη στήσω. Άρα πρέπει μετά να υπάρχει δυνατότητα να υποστηριχθεί αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα και σε επίπεδο οικονομικό ακόμη και κοινωνικό. Και σε αυτό θέλω να σταθώ, ότι προσπαθούμε να έχουμε καλύτερη συνεννόηση στην κοινή μας στόχευση και να αντιληφθούμε ότι συμβάλλουμε στη σταθεροποίηση και στη σταθερότητα στη γειτονία μας. Η Λιβύη, επί παραδείγματι. Μη κυβερνητικέ οργανώσεις που έχουν αναλάβει από εμά ε, εκτέλεση έργων για λόγους ασφαλείας δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να απορροφήσουν και να διαθέσουν τα κονδύλια που έχουμε έτοιμα. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει ακόμα και αυτό να το διακινδυνεύσουμε. Διότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λιβύη είναι απαράδεκτη και αν δεν έχουμε επιτυχία, η αποτυχία μας θα, θα φέρει και πολύ γρήγορα αποτελέσματα δυσμενή για μας. Η μετανάστευση που θα περάσει και από τη Λιβύη είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και τις εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπιστέντες, Λιβύους πολίτες, που λόγω της ε, οικονομικής, ε, πολιτικής αλλά πάνω απ' όλα κατάστασης της ασφάλειας στη χώρα είναι υποχρεωμένοι να καταλήψουν τις αιστείες τους και να μετακινηθούν εσωτερικά έστω μέσα στη χώρα. Πρέπει ταυτόχρονα λοιπόν να κοιτάξουμε και αυτή την διάσταση και να ε, κοιτάμε και τα κονδύλια να διατίθενται σωστά αλλά και να φτάνουν στον τελικό αποδέκτη. Αλλά ταυτόχρονα βρισκόμαστε και αντιμέτωποι με την αδυναμία να επαληθεύσουμε τα γεγονότα αυτά. Και πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε διαφορετικές απόπειρες ή δοκιμές. Είναι η πραγματικότητα που μας φέρει αντιμέτωπους με αυτές τις συνθήκες. Παραδείγματι, στην πρόσφατη ιστορία, στη γειτονία της Ευρώπης, δεν υπάρχει ε, προηγούμενο κράτους που να ε, έχει μείνει χωρίς πολιτική ηγεσία για χρόνια όπως η Λιβύη. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα το ε, αντιμετωπίσουμε αυτό. Εγώ δεν έχω να σας δώσω καμιά μαγική συνταγή. Απευθύνω όμως έκκληση να διατηρήσουμε ευελιξία και πνεύμα ε, ε, ανοιχτό, ώστε να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε διαφορετικές λύσεις και να δούμε αν μια από αυτές φέρνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Χωρίς όμως να μπορώ να εγγυηθώ ότι κάθε μέτρο που θα αναλάβω θα φέρει την επιτυχία. Απλώ ξέρω πολύ καλά ότι θα ήταν λάθος να μην πράξουμε τίποτα. Γιατί εκεί σίγουρα θα έχουμε αποτύχει. Το ότι κάθε μέτρο που θα υλοποιήσουμε ή θα προτείνουμε θα φέρει σε χώρες όπως η Συρία σε χώρε οπως η Λιβύη τα αναμενόμενα ε, και επιθυμητά αποτελέσματα, όχι, δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Κύριε Τσόφκο. Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ Επίτροπε, θα είμαι σύντομη γιατί είναι πολύ αργά και έχετε ήδη μιλήσει πολύ απόψε. Πρόσφατα η Επιτροπή ΑΦΕΤ στην γνωμοδότησή της εξέφρασε ανησυχία σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν για μείωση του μέσου του για προενταξιακή αρρωγή προς τα Δυτικά Βαλκάνια και την μείωση κατά 90 εκατομμύρια ευρώ του συγκεκριμένου κονδυλίου. Μπορείτε να μου εξηγήσετε αν θα το κάνετε κάτι γι' αυτό, αν θα επανεξετάσετε αυτή την πρόταση. διότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων ε, στο διοικητικό επίπεδο και στο, όσον αφορά το κράτος δικαίου για αυτές τις χώρες που προσδοκούν στην προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ημέρα των ημερών. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση σας και επίσης να καλωσορίσω τα όσα μας είπατε για την ανάγκη να δοθεί περισσότερη ορατότητα στις ευρωπαϊκές χώρες να συνεχιστεί η διεύρυνση ώστε να υπάρχει σταθερότητα και ειρήνη στα σύνορα. Οπότε είναι απαραίτητη μια διπλωματία όσον αφορά τα, τις βαλκανικές χώρες και εγώ θα ήθελα να συνεχίσετε σε αυτή την ε, πορεία γιατί είναι ένα σημαντικό μέσο διπλωματικό το οποίο δεν χρησιμοποιεί όπως δει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Στην ε, διάμεση μας ε, έκθεση πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατότητες των υποψηφίων χωρών και αυτό το έχουμε συζητήσει και από διάφορες απόψεις και σήμερα ότι αν υπάρχει δηλαδή έλλειψη δυνατότητας απορρόφησης, αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα ποσά τα οποία βάζουμε στον προϋπολογισμό ή, εν πάση περιπτώσει, χορηγούμε στην κάθε χώρα. Αλλά στόχος, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι να ξεκονομήσω χρήματα, αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα αυτά δαπανώνται σωστά. Εάν κανείς εξετάσει όλες τις χώρες, θα δει πόσα project υπάρχουν και πόσα χρήματα χορηγούνται σε κάθε χώρα. Αν μια χώρα δεν μπορεί να τα απορροφήσει, τότε προσπαθούμε να τα μετακινήσουμε σε μια άλλη. Και είναι ένας από, από το στρόπους αναγνώρισης των πορισμάτων μας, δηλαδή μάλλον της, της δράσης μας, ότι πολλές φορές ήμασταν εξαιρετικά φιλόδοξοι στο παρελθόν για να μεταφέρουμε τις διαχειριστικές αρμοδιότητες και ευθύνη προς τα υποψήφιες χώρες ενώ από ό,τι φάνηκε έπειτα δεν ήταν αρκετά προετοιμασμένες και όριμες και γι' αυτό και αποφασίσαμε να εφαρμόζουμε περισσότερη άμεση διαχείριση από ό,τι στο παρελθόν, έτσι ώστε να εγγυηθούμε την ορθή εφαρμογή. Αλλά επίσης, πρόθεση τότε για μεταφορά των ευθυνών προς τις υποψήφιες χώρες για ώστε να διαχειριστούν τα χρήματα δηλαδή μόνες τους την εμπνευστήκαμε από την πρόθεσή μας να είναι καλά προετοιμασμένα για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα διευθυντικά ταμεία ε, οι χώρες αυτές. Αλλά και πάλι από ό,τι φάνηκε ήμασταν εξαιρετικά φιλόδοξοι και πρέπει να εξισορροπήσουμε εκ νέου τον τρόπο με τον οποίο ε, παρέχουμε χρήματα, πώς αυτά χρησιμοποιούνται, ώστε να έχουμε τα απαραίτητα project, αλλά να εφαρμόζονται, αλλά να έχουμε και την απαραίτητη στήριξη για τις μεταρρυθμίσεις είναι ένα από τα παραδείγματα που πρέπει ναι, να σταθμίσουμε εκ νέου την πολιτική μας και την προσέγγιση μας. Αλλά και πάλι να πω ότι κάθε υποψήφια χώρα θα πρέπει να μπορέσει να σταθεί ικανή, να διαχειριστεί τα του οίκου της με βάση όμως σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει στο τέλος αυτής της βραδιάς να μιλήσουμε για την Τουρκία. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί δέχεται πολλά χρήματα. Πρώτη μου ερώτηση λοιπόν. Πώς αναπτύσσεται αυτή η κατανομή των κονδυλίων μετά την επίσκεψή μας είχαμε την εντύπωση ότι ε, θα έπρεπε να επιστρέφεται ολόκληρη η προενταξιακή βοήθεια. Δεν συμβαίνει όμως αυτό που αυτό μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς ε, αξιοποιείται σε τελευταία ανάλυση αυτή η προενταξιακή βοήθεια γιατί η Τουρκία εξελίσσεται σε ένα κράτος το οποίο όλο και, όλο και απομακρύνεται από την ένταξη. Τι νόημα λοιπόν έχει, σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι χρήσιμη αυτή η προενταξιακή βοήθεια. Μήπω λοιπόν αντί να μιλούμε για διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων πρέπει να κοιτάξουμε να ε, σταματήσουμε την ε, καταβολή της ε, προενταξιακής βοήθειας. Δεν βλέπουμε ότι ριζοσπαστικοποιείται διαρκώ και η δημόσια διοίκηση της Τουρκίας. Δεν έχετε ανησυχία για τα κονδύλια τα οποία διοχετεύονται σε σημεία της διοίκηση που δεν είναι πλέον ορατό σε ποιον πηγαίνουν και μήπω πηγαίνουν και σε ανθρώπους ριζοσπαστικοποιημένους απάντηση για την κυρία Γκρέσλη για να απαντήσω στην πρώτη σας ερώτηση. Της περαιτέρω διάθεση της πρωταξιακής βοήθειας η απάντηση είναι ότι την απόφαση αυτή, την, η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε πολιτικό επίπεδο. Θα μπορούσε να αποσυνδεθεί βεβαίως νομικά, αλλά να ανακτηθεί, να μειωθεί ή και να σταματήσει η αναπτυξιακή βοήθεια, η προενταξιακή βοήθεια, θα ήταν αντίθετη με τα κριτήρια κράτους δικαίου και τα λοιπά. Ε, τα νομικά κριτήρια. Διότι αν το πράταμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε και τα κράτη-μέλη μας να υποστούν αντίστοιχη, θα υφίσταν το και τα κράτη-μέλη αντίστοιχη πίεση Εάν περικόπταμε δηλαδή, σταματούσαμε την παροχή της προταξιακής βοήθειας λέγοντας ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Τουρκία ενώ ταυτόχρονα ενώ ε, ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Τουρκία, συνεχίζουμε τουλάχιστον σε νομικούς όρους τις διαπραγματεύσεις, ε, είναι οξύμορο και άρα θα πρέπει να γίνει μια πολιτική κατά κύριο λόγο αξιολόγηση κοινή αξιολόγηση. Πιστεύω ότι έχει προκύψει σχετική δυναμική βεβαίως, η προοπτική αυτή, αλλά ταυτόχρονα και το είδαμε στο Ταλίν, στον Κιμνίχ, θα πω ότι η θεώρηση που έχουν τα κράτη-μέλη προς Τουρκία είναι διαφορετική, δηλαδή υπάρχουν κράτη, Γερμανία, Αυστρία, αλλά και κάποια άλλα, όχι πολλά όμως, που έχουν διαφορετικές ευαισθησίες. Διότι έχουν ε, μειονότητα τουρκική, λέει ο μιλητής. Και βέβαια αντιμετωπίζουν ε, και τις ε, πιέσεις, δηλώσεις, επιθέσεις από πλευράς της Τουρκίας. Λεκτικές επιθέσεις. Άλλες χώρες που δεν έχουν τουρκική μειονότητα έχουν ε, ίσως διαφορετική θεώρηση, γεωστρατηγική θεώρηση. Ε, μπορεί να παίζει διαφορετικό ρόλο για αυτά τα κράτη η Τουρκία. Η Τουρκία είναι ταυτόχρονα και μέλος του ΝΑΤΟ, άρα έχουμε να κάνουμε με, με ένα πεδίο δύσκολο και σε επίπεδο γεωστρατηγικό και γεωπαθητικό. Άρα δεν είναι ότι αφήνουμε να μας εκβιάζουν, ε, ή όπως αλλιώς θα το πει κανείς, αλλά ότι βλέπουμε διαφορετικά στοιχεία χαρακτηριστικά, διαφορετικές ε, ε, πτυχές του ζητήματος και βεβαίως ε, οι απολύσεις, ε, συλλήψεις, φυλακίσεις χιλιάδων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στην Τουρκία ασφαλώς και έχουν συνέπειες ως προς την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης ίσως όχι στο βαθμό που θα μπορούσε κανεί να περιμένει. Δεν είναι δηλαδή τόσο τραγικά τα πράγματα. Αλλά η Τουρκία είχε πάντοτε προβλήματα απορροφητικότητα των κονδυλίων. Αυτό πρέπει να το καταγράψουμε στην μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Και έχω τώρα προχωρήσει σε μέτρα όπου σταματούν ορισμένα προγράμματα στο χώρο της δικαιοσύνης όπου δεν έχουμε εγγύησεις για το πώς θα αξιοποιηθούν τα μέσα αυτά. Είχαμε κάνει τα τελευταία χρόνια προσπάθειες και δαπανίσει κονδύλια για την κατάρτιση δικαστών επί παραδείγματι άλλων λειτουργών της δικαιοσύνης και μάθαμε ότι το μεταξύ αυτοί απολύθηκαν. Πού πήγαν τα χρήματα λοιπόν αυτά. Ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε να αντιστρατευτούμε αυτές, δεν μπορούμε να ανατρέψουμε αυτές τις εξελίξεις. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να πατήσουμε το φρένο κινδύνου θα έλεγα. Ε, ταυτόχρονα δεν μπορούμε και να εγκαταλείψουμε τον, ε, τους πολίτες Τουρκίας ε, που και στο τελευταίο δημοψήφισμα κατά 50% είχε κάνει, είχαν κάνει διαφορετικές επιλογές. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ο Ερντογάν είναι η Τουρκία. Ο Ερντογάν είναι πρόεδρος, ε, το ΑΚΠ είναι το κυβερνών κόμμα βεβαίως, αλλά το ίδιο το δημοψήφισμα, το πρόσφατο δημοψήφισμα απέδειξε ότι υπάρχει σημαντική, σημαντικό ρήγμα στον πληθυσμό και γι' αυτό καλό θα ήταν να διατηρήσουμε τις επαφές, το διάλογο, τη συνομιλία με τη χώρα, με τους πολίτες της, ώστε να μην στραφεί εναντίον μας αυτή, αυτή η κατάσταση. Και δεν μιλώ για πρόσφυγες τρίτων κρατών, αλλά για πρόσφυγες Τούρκους. Άρα λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε και να τακτοποιήσουμε, να συγκυρίσουμε τα πράγματα και να επαγρυπνούμε ώστε να αξιοποιούνται σωστά τα κονδύλια και βεβαίως η πρόθεσή μας είναι να ε, είμαστε πάντα πάρα πολύ προσεκτικοί ως προς τα χρήματα τα οποία ε, διαθέτουμε και τον τρόπο με τον οποίο αυτά αξιοποιούνται. Κύριο Σπίξτα, το ελεκτικό συνέδριο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα πρέπει να πω ότι ήταν η συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ε, και από την πλευρά των Ευρωβουλευτών και από την πλευρά του Επιτρόπου και χαίρομαι που μπόρεσα να έρθω σε αυτή τη συνεδρίαση με τη, διότι είχαμε πολλή δουλειά το απόγευμα και αύριο επίσης. Ε, ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η συζήτηση. Ε, είναι ικανοποιητικό να ακούει κανείς ότι τα, οι εκθέσεις μας διαβάζονται παρόλο ε, που ε, για την Επιτροπή ε, ε, πάντα το ποτήρι είναι μισό γεμάτο ενώ για τους ευρωβουλευτές άδειο. Πέρσι είχαμε έξι εκθέσεις, τρεις για την Επιτροπή Γειτονίας και τρεις για την ένταξη. Και είχαμε την έκθεση για την, την Ισία. Στις 26 Ιουνίου είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και χαίρομαι που επέσυρε την προσοχή των μελών αυτές της Επιτροπής. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία. Διαβαστήκανε όλα τα έγγραφα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία υπό το φως των απαντήσεων του κυρίου Επιτρόπου. Θα βρείτε στις εκθέσεις ότι πάρα πολύ συχνά υπάρχει έλλειψη δέσμευσης από την πλευρά των δικαιούχων. Αυτές οι χώρες λαμβάνουν τεράστια κονδύλια των φορολογουμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα υπάρχει έλλειψη δέσμευσης. Αυτό οδηγεί στο σημείο που ανέφερε ο Επίτροπος των κινήτρων των κινήτρων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή ή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πίεση ελαφρά ή βαρύτερη από πλευρά της Κομισιό. Υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτίωσης. Ο Επίτροπος Χαν μίλησε για μόχλευση ε, περισσότερες φορές από μία. Και νομίζω ότι είναι μια ιδέα πολύ ενδιαφέρουσα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, χρησιμοποιήσει την επίδραση που έχει, την, ε, την πίεση, τη δύναμη πίεσης που έχει για να ξοδεύονται καλά τα χρήματα. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους για το πώς μπορούμε να ε, ευελτιώσουμε αυτήν την πίεση από επίδραση από πλευράς των φορολογουμένων. Επίσης μιλήσατε για διαφάνεια. Είναι καλή η πρόταση. Θα πρέπει να γίνουν τα πράγματα πιο διαφανή και να είμαστε σαφείς όταν ξοδεύουμε χρήματα σε μια χώρα της γειτονίας ή σε χώρα υποψήφια να να πούμε ακριβώς στους Ευρωπαίους πολίτες ποιοι είναι οι στόχοι που πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι. Αυτά είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται, ποια είναι τα benchmark, τα σημεία αναφοράς, ποια έχουν επιτευχθεί, ποια δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί για το πώς ξοδεύονται τα χρήματα συνδέοντας τους εαυτούς μας και συνδέοντας την Επιτροπή με στόχος, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία θα μπορούμε να ασκήσουμε ε, περισσότερη πίεση δίνοντας κίνητρα ε, στους δικαιούχους. Δεύτερο ε, σημείο είναι η σημασία της ΤΕΦΑ. Η ΤΕΦΑ είναι μια ένδειξη για το πώς και σε ποιο βαθμό το δημόσιο <coughs> χρήμα που δίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τύχει χρηστής διαχείρισης, δημόσιας χρηστής διαχείριση. Όπως γράφουμε στην έκθεση για την Τινησία, η ε, ΠΕΦΑ ε, θα πρέπει να ε, μας επιτρέπει να αξιολογούμε καλά τα πράγματα. Είναι πάνω από 7 χρόνια τώρα. Νομίζω ότι υπάρχει καλός λόγος γι' αυτό, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τα δημόσιο χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ξοδεύεται καλά και θα πρέπει να βεβαιωνόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο ότι ξοδεύεται καλά ε, και ότι έχουμε ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην περίπτωση της Τινησίας υπάρχει, υπήρχε κάποιο περιθώριο βελτίωσης για να πούμε τα πράγματα αρκετά ήπια. Ευχαριστώ και πάλι για, για την πάρα πολύ σημαντική συζήτηση. Ευχαριστώ όλα τα μέλη που συμμετείχαν εδώ. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε εσάς κύριε Επίτροπε. Πάνω από δύο ώρες ήσασταν στη διάθεσή μας. Είμαστε πάντα στο πλευρό σας, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι το έργο σας. Δεν σταματούμε βεβαίως. Θα προσπαθούμε πάντοτε μαζί σας για καλύτερα αποτελέσματα. Και σας διαβεβαιώ ότι αν μπορούσαμε να ασκήσουμε και περισσότερες πιέσεις θα το είχαμε πιέσει. Έχει περάσει η ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και θα ξανασυντηθούμε στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις 25 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή νύχτα. Πέρα συνεδριάσεως.